Ξεκινούμε τη συνεδρίαση, λέει η Πρόεδρος. Ραμόν, κάτσε κάτω. Ε, Σε ευχαριστώ. Άρχισε η συνεδρίαση και σα ενημερώνω ότι μεταδίδεται στο ίντερνετ τη συνεδρίασή μας. Πάμε στο πρώτο θέμα που είναι η έγκριση της ημέρησας διάταξης σας έχει διανεμηθεί στις 21 Νοεμβρίου και θα πρέπει να σας πω για δύο αλλαγές που έχουν γίνει. Πρώτα πρώτα υπάρχει ένα αίτημα του Αλέν Λαμασούρ, το σχέδιο εκθεσής του όσον αφορά την αναβαθμισμένη συνεργασία που ήταν το 8 διατάξει συνθήκων για ενισχυμένη συνεργασία θα συζητηθεί στις 10 και 4 νωρίτερα. Οπότε και οι ψηφοφορίες αντίστοιχα θα γίνουν πιο αργά. Οπότε παρακαλώ ενημερώστε οι βοηθοί τους βουλευτές, ότι έχει πει η γραμματεία ήδη με email και επίσης άλλη αλλαγή το 12 η συνεδρίαση με τον Μπαρνιέ και το επιτελείο του θα γίνει στις 4 και θα πρέπει να φύγει στις 5 και θα συνεχίσουμε μετά μέχρι τις 5.30 τη συζήτηση με τους ε, συναδέλφους. Θα γίνει και κλεισμένο θυρών αυτή η συνεδρίαση. Αν δεν έχετε τώρα κάποια αντίρρηση, θεωρώ ότι εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε η μέσα διάταξη όσον αφορά τώρα τις ανακοινώσει μου που είναι το δεύτερο σημείο της μέσα διάταξης είναι το ότι για τεχνικούς λόγους Οι τροπολογίες για την έκθεση για τον διομεσολαβητή θα είναι μόνο στα αγγλικά. Τα άλλα ισχύουν αυτό γιατί έτσι μας είπε η υπηρεσία μετάφρασης. Έχουμε επίσης την Ολομέλεια της Κοζάκ στην ε, Βιέννη. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, και ήμουν συμπρόεδρος με την κυρία Μαγκίνες, τον κύριο Ροντρίγκε. Επίσης είχαμε τον Οτμαρ Κάρας ε, ως Αυστριακό και επίσης παρακολούθησαν τις εργασίες μας και κάποιοι Αυστριακοί άλλοι ε, ευρωβουλευτές. Επίσης ε, είχαμε και βουλευτές του Εθνικού Κοινοβουλίου της χώρας, ε, ενδιαφέρουσες ζωντανές συζητήσεις. Επίσης μίλησα και στη θέση του κυρίου Μπαρνιέ, ο οποίος ήταν επισχολημένος στις διαπραγματεύσεις του Brexit. Ενημέρωσα για αυτή την υπόθεση. Επίσης ε, από το Βρετανικό Κοινοβούλιο είχαμε τον ε, William Cash ε, που είναι υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου επίσης η Μέρη Μαγκίνες ε, που είναι η υπεύθυνη για τη σχέση με τα Εθνικά Κοινοβούλια εκείνη μίλησε για ε, τα θέματα διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν αξιόλογη αυτή η συνεδρίαση γιατί είδαμε ότι υπάρχει σύγκληση απόψεων ε, όσον αφορά το Brexit. Επίσης, προέκυψε αυτό το γνωστό ότι λυπούμεθα που αποχωρεί το Μέρο Βασίλειο, αλλά σεβόμαστε την αποφασή τους. Αυτά όσον αφορά την Βιέννη και επίσης ε, είπαμε ε, τα των ευρωεκλογών τώρα όσον αφορά τις προτάσεις των συντονιστών αποφάσισαν κάτι που έχει σχέση με τις εργασίες μας Έχουμε γνωμοδότηση σε σχέση με την έκθεση της ε, Νομικής Επιτροπής για την ετήσια έκθεση της Επιτροπής του 17 όσον αφορά την αναλογικότητα και την επικουρικότητα. Θα την αναλάβει το ΕΛΚ και συγκεκριμένα ο Έλμαρ Μπροκ. Αν δεν έχετε ενστάσεις, θεωρώ ότι εγκρίνεται η απόφαση αυτή των συντονιστών. Επίσης, Ε, έχουμε τα πρακτικά τη συνεδρία της 24 η του Μαΐου και αν δεν υπάρχει ένσταση και αυτά θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Αυτό θα γίνει αν δεν έχουμε ένσταση μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Οπότε και προχωρούμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 5. Είναι η δεύτερη φορά που η ΑΦΚΟ οργανώνει αυτή την εκδήλωση για την νεολαία, το ΆΙ. Έγινε το ίδιο και το 16 τον Αύριο. Επίσης είχαμε μια εκδήλωση κατά την σύνοδο του Ιουνίου στο Στρασβούργο. Ισχύει αυτή η εκδήλωση υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια και θα ακούσουμε από εσάς τώρα πώς αξιολογείται ε, αυτή την εκδήλωση που εμείς διοργανώνουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία επομένω να ακούσουμε τους νέους που ήρθαν να ακούσουμε τη γνώμη τους για το μέλλον της ε, Ευρώπης να μας πείτε τι θεωρείτε ότι είναι τα πιο σημαντικά, τι όνειρα έχετε, τι ιδέες έχετε σε σχέση με την δική μας δουλειά. Σας έχουμε διαβάσει ένα κείμενο με συγκεκριμένες ε, προτάσεις, συνάδελφε, για εκείνη την συνάντηση στο Στρασβούργο. Συντάξαμε και κάποια έκθεση και ε, σε άλλες επιτροπές επίσης ε, προσκαλούμε τους νέους έχουμε αυτή τη φορά 7 κοινοβουλευτικές επιτροπές Οκτώβριο και Νοέμβριο που ασχολούνται σε κάποιες κοινέ συνεδριάσεις με τους νέους. Ακούσουμε τι σας απασχολεί, πολύ σημαντικό Επίσης να δούμε πώς βλέπετε το μέλλον της Ευρώπης μετά το Brexit, την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, την συμμετοχή στις ε, ευρωεκλογές και πως η Ευρώπη θα είναι ένα αυθεντικό βήμα συζήτησης όλα όσα θα μας πείτε θα είναι ενδιαφέροντα. Έχουμε εδώ τρεις συναδέλφους. Ε, ξεκινάμε με τον Ανδρέα που προέρχεται από την Μακεδονία. Επίσης τον Καλογιαν Χοφμάιστερ, που είναι βούλγορο-γερμανός. Μισός Γερμανός, μισός ε, Βούλγαρος και τον ε, Άντρα Σνάγκη από την Ουγγαρία. Μιλήσουμε για τους τρεις θεματικούς μας άξονες και κατόπιν ε, οι συνάδελφοι της Επιτροπής θα τοποθετηθούν για τόσα εσείς έχετε να μας πείτε. Πρώτα πρώτα ξεκινούμε με το ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης μετά το Brexit. Ανδρέα, εσύ πάρει πρώτο στην ε, σκητάλη. Πόση ώρα έχετε... Α, δύο λεπτά, δύο λεπτά. Έτσι προβλέπετε εδώ στο κοινοβούλιο. Στην Ολομέλεια συνήθως ε, μιλάμε ένα, ένα. μισή, δύο λεπτά. Τέλος πάντων, ε, αυτό είναι μια πρόκληση για σας. και μετά θα σχολιάσουν οι συνάδελφοι. Ανδρέα. Η Ανδρέα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, καλημέρα στα μέλη της Επιτροπής ΑΦΚΟ. Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας ε, μοιραστώ μαζί σας κάποιες ιδέες που προέκυψαν από την ε, εκδήλωση νεολαίας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες της εκπαιδευτικής και κινητικότητας μετά από τον Brexit. Το Brexit είναι μια λέξη η οποία μας έχει ήδη κουράσει όλους, δηλαδή έχουμε κουραστεί να την ακούμε, ε, νομίζω όλοι θα συμφωνήσετε, αλλά έχει το δυναμικό να επηρεάσει πάρα πολύ τις ε, ζωές ε, πολλών ανθρώπων και δεν αποτελεί βέβαια το ότι ένας σημαντικός αριθμός workshop έλαβε χώρα μόλις ανακοινώθηκε το Brexit και χαίρομαι που υπάρχουν πολλοί νέοι που συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για να υπάρχουν οι αμοιβέ ανταλλαγές στον εκπαιδευτικό τομέα. και χαίρομαι πολύ που έχω τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω κάποιες από αυτές τις ιδέες. Η Δυνατότητε αυτέ, οι εκπαιδευτικέ και δυνατότητες, ε, ε, οι ευκαιρίες ε, κινητικότητα μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο μετά τον Brexit, αλλά θα πρέπει να τι διατηρήσουμε. Γιατί οι νέοι θα πρέπει να έχουν τι ίδιε ευκαιρίε σε ό,τι αφορά την προσωπική του ανάπτυξη και τον διαπολιτισμικό διάλογο, όπω και οι γενιέ πριν από αυτού. Δηλαδή, εάν χάσουν την πρόσβασή του σε προγράμματα όπω το Erasmus Plus και το EVS, δεν θα έχουν τη δυνατότητα πλέον να προβαίνουν σε ανταλλαγέ με άλλου φοιτητέ και σπουδαστέ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ λοιπόν πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παραμείνει μέσα στο Erasmus σε, διασφαλίζοντας έτσι τις ανταλλαγές φοιτητών και σε ταμικό και σε συλλογικό επίπεδο. Και θα ήθελα επίσης το ΕΒ να συνεχίσει να συμμετέχει στο διαστρωμένο διάλογο ε, έτσι ώστε να μπορούν και οι νέοι να έχουν και κάποιο λόγο στην μετά τον Brexit εποχή. Επίσης, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο ζήτημα των θεωρήσεων. Ε, αποτελούν οι θεωρήσεις ένα διοικητικό και οικονομικό άκτος για τους ε, ανθρώπους, οπότε αν τους επιβληθούν θα περιορίσουν την κινητικότητά τους και θα επηρεάσουν τις διαπολιτισμικές τους ε, σχέσει. Πιστεύω πω οι νέοι δεν θα πρέπει να έχουν λιγότερες ε, δυνατότητες και ευκαιρίες ε, εκπαίδευσης και κινητικότητας ε, απλώς και μόνο επειδή υπάρχει ένα πολιτικό αδιέξοδο. Οπότε θα ήθελα να καλέσω εσάς τα μέλη της ΑΦΚΟ να διασφαλίσετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμένει στο Erasmus Plus και ότι θα παραμείνει και μέσα στον διαδρομένο διάλογο για την νεολαία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εδώ μεταξύ έχω αναλάβει την Προεδρία και λογαριασμό της κυρίας Ούμπνερ, γιατί με το αρχαιότερο μέλος εδώ. έχετε να παρουσιάσετε και μια δεύτερη ιδέα, οπότε συνεχίστε παρακαλώ. Η δεύτερη ιδέα που θα ήθελα να σας παρουσιάσω είναι οι ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια του Brexit, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις νέες ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προκύψουν. Παρά δηλαδή τις προκλήσεις που δημιουργεί το Brexit, δημιουργεί και δυναμικό σε ό,τι αφορά τις αλλαγές και τις βελτιώσεις. Αποτελεί λοιπόν μια ευκαιρία βελτίωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και προκειμένου να έρθει σε επαφή περισσότερο με τους ανθρώπους στις, ε, ε, περιοχές, στις αγροτικές περιοχές με έναν τρόπο ο οποίος έχει περισσότερο νόημα. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παίξει ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά το δημοκρατικό ενδιαφέρον των νέων, ε, καθώ μπορεί να το κάνει σε ορισμένε περιπτώσει καλύτερα και από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Μπορεί δηλαδή να επιτρέψει άμεση, ε, άμεσο δικαίωμα ε, ψήφου, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά του επιτρόπους και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να συνεισφέρει σε μια πιο δημοκρατική Ευρώπη. Ε, ενδεχομένως να υπάρχει και περισσότερη αίσθηση ούτως ώστε να αυξηθούν οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποτελεί και το μόνο άμεσα αρετό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές οι περισσότερες εξουσίες θα μπορούσαν για παράδειγμα ε, να συμπεριλαμβάνουν την υιοθέτηση περισσότερων εκθέσεων ε, και ψηφισμάτων. Προφανώς το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα περισσότερο από ποτέ θα συνεχίσει να αποτελεί ζήτημα προτεραιότητες. Οπότε ε, μία ακόμα ευκαιρία κατά τις επόμενες ευρωεκλογέ θα μπορούσε να είναι η δημιουργία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο ε, μιας επιτροπής η οποία θα ασχολείται ειδικότερα με το μέλλον των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα μπορούσε να αφουγκράζεται αν θέλετε τους και να παρακολουθεί τις ιδέες τους καθώς γίνονται οι νέες συστάσεις στο πλαίσιο του διαθρομένου διαλόγου. Ε, θεωρώ πως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς το να καταδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ενδιαφέρεται για τους νέους της. Νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που δίνει το Brexit, ούτως ώστε να δώσει ε, περισσότερη πρόσβαση και να είναι πιο ανοιχτή απέναντι στους νέους και προκειμένου να θίξει τα ζητήματα που τους αφορούν ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, τα μέλη τώρα της Επιτροπής μπορούν να παρέμβουν, να το επιθυμούν. Ραμόν, λοιπόν, έχει ζητήσει πρώτος το λόγο. In which case, uh, let me say a few things, but then the floor is definitely back to you whenever you're ready. Um, basically, my... Uh... Επιτρέψτε μου να θέσω εγώ τότε ένα ερώτημα. Και εγώ λυπάμαι φυσικά για το Brexit. Αλλά θεωρώ πως είναι σωστό που το αντιμετωπίζετε και ως ευκαιρία. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω ένα κλισέ, αλλά νομίζω πως αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να ε, ξανασκεφτούμε λίγο τι ακριβώς ε, κάνουμε ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω ε, είναι γιατί θεωρείτε πως οι νέοι άνθρωποι έχουν καλύτερες ιδέες από ότι μεγαλύτερη σε ηλικία άνθρωποι. Γιατί ορισμένε ε, φορέ έχουν πράγματι καλύτερε ιδέε οι αλλά ορισμένε φορέ όχι. Οπότε πώ ε, μπορείτε να φιλτράρετε, αν θέλετε, να δεθείστε τι καλέ ιδέε των νέων. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι σε σχέση με αυτές τις ευκαιρίες που δημιουργεί το Brexit είναι τι έχει επιτύχει το Brexit σε ό,τι αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όλοι νομίζω πως είμαστε πλέον βέβαιοι ότι θα λάβει η χώρα το Brexit, δηλαδή 19 Μαρτίου. Αλλά τι θα επιτύχει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να μην συμφωνήσετε μαζί μου, αλλά εγώ θεωρώ πως στο πλαίσιο του Brexit τα ε, ε, υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη έχουν επιδείξει μια πρωτόγνωρη ενότητα. Τι θεωρείτε εσείς από την πλευρά σας. Θα μιλήσω ισπανικά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακούμε την νεολαία ιδίω σε ένα τέτοιο δομημένο πλαίσιο και μετά και τις συνεδριάσεις ε, που έχουν πραγματοποιηθεί. Το δικό μου ερώτημα είναι το εξής. Βλέπετε εσείς σε διάφορες ε, χώρες ε, η νεολαία να έχει διαφορετικές γνώμες για την Ευρώπη. Όταν απευθύνεστε σε όλους αυτούς τους νέους με τους οποίους μιλάτε, έχουν την ίδια στάση, τον ίδιο ενθουσιασμό απέναντι στο μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύετε ότι όλοι έχουν, λοιπόν, ε, βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Οι νέοι των ευρωπαϊκών χωρών έχουν την ίδια στάση. Και μετά μιλήσετε για αυτό το πάθος ε, που μας κινεί προς ε, το μέλλον της Ευρώπης, αλλά Τις προηγούμενες δεκαετίες εμείς τότε μιλούσαμε και είχαμε στο νου μας ε, το ευρωπαϊκό όραμα ως έναν χώρο ειρήνης λόγω του πολέμου προηγουμένως και έναν χώρο ευημερία. Ίσως για τους νέους σήμερα η ειρήνη να είναι κάτι το δεδομένο στη ζωή τους. Επομένω, κατέχει την ίδια βαρύνουσα σημασία η ειρήνη όπως είχε για τότε και για την πρόοδο. Ε, για εμάς υπήρχε πάντα μια θετική και ανωδική πορεία, ενώ για σας το μέλλον είναι αβέβαιο. τα ύδατα. Και όταν ε, σκέφτεστε το μέλλον της Ευρώπης, τι είναι αυτό που πραγματικά σας κινητοποιεί Τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι το μέλλον της Ευρώπης είναι σημαντικό. Ευχαριστώ. Helmut. you, Ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια που άκουσα. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και τους δυο σας και ήμουνα και το Μάιο σε αυτή την εκδήλωση. Μιλήσατε για το Brexit και οι δύο και είπατε ότι θα πρέπει να εμπλέξουμε περισσότερο τους νέους ε, στην ε, διαδικασία λήψης πολιτικής. Το θέμα είναι γιατί οι νέοι όμως δεν συμμετείχαν στο δημοψήφισμα για ένα θέμα που θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει εξαιρετικά, ε, γιατί όλοι κατανοείτε και γνώριζαν μάλλον τη σημασία του δημοψηφίσματος. θέλουν λοιπόν την συμμετοχή των νέων ε, στην διαδικασία λήψη πολιτικής. Αλλά πλέον αυτό δεν είναι τόσο προφανές, γιατί όλοι τα θεωρούν όλα δεδομένα. Τι θεωρείτε λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουμε ε, στην επικοινωνία μας με τους νέους, για να τους πλησιάσουμε περισσότερο και να τους πείσουμε να συμμετάσχουν στα κοινά. Ευχαριστώ. Μάιτα. Ευχαριστώ, θα μιλήσω ισπανικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Είστε Ευρωπαίοι πολίτες. Θα ήθελα όμως να μου πείτε τι θεωρείτε ότι ενέχει αυτή η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τους νέους ως Ευρωπαίους πολίτες. Στην ΑΦΚΟ εξετάζουμε διάφορες επιτροπές που αναφέρονται ακριβώς σε αυτό το ζήτημα, γιατί υπάρχει η πεποίθησή μας, η αντίληψή μας και μετά υπάρχει και η πραγματικότητα. Και μεταξύ των δύο πολλές φορές υπάρχει μεγάλο χάσμα. Επειδή είστε τόσο νέοι, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Ποια θεωρείτε λοιπόν ότι είναι τα πραγματικά χαρακτηριστικά ε, της ευρωπαϊκής ε, ηθαγένειας και απονομική σκοπιά, σκοπιάς. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό για να καλύψουμε τυχόν κενά. Ευχαριστούμε για αυτά τα ερωτήματα. Δίνω τώρα το λόγο στην Αντρέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πολύ προσφύγει όλα τα ερωτήματα και σας ευχαριστώ που μου τα θέσατε και ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω σε όλα αυτά γιατί δεν είμαι και εγώ εμπειρογνώμων προς το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν το ήξερα βέβαια θα ασχολούμουν με αυτό περισσότερο. Αλλά επιτρέψτε μου λίγο να αναφερθώ καταρχήν σε ό,τι αφορά την, την πρόοδο, σε ό,τι αφορά την περισσότερη Ευρώπη. Καταρχήν, ε, γιατί οι νέοι, με ρωτήσατε, έχουν καλύτερε ιδέε από τη μεγαλύτερη ηλικία. Εγώ στην ε, εργασία μου ε, έχω συνέχεια επαφή με νέου θεωρώ πω όταν γίνεται η δίνεται περισσότερη εξουσία ε, σε ζητήματα που τους αφορούν πράγματι ε, μπορούν να συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό. Ε, και έχουν ενδιαφέρουσες ιδέες γιατί υπάρχει ένα σαφές χάσμα γενναιών όπως αναφέρθηκε. Δηλαδή υπάρχει μια γενιά ευρωβουλευτών ε, οι οποίοι μεγάλωσαν ακόμα με τον πόλεμο και εκτιμούν πολύ ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αποτέλεσε ένα project, αν θέλετε, ειρηνευτικό. Αλλά υπάρχει τώρα, ε, υπάρχουν οι νέε γενιέ, οι οποίε είχαν το προνόμιο του να γεννηθούν στην ειρήνη και κατά συνέπεια θεωρούν το ναι, την Ευρωπαϊκή Ένωση ω ε, κάτι το δεδομένο. Άρα λοιπόν αυτό θεωρώ πώ έκανε το Brexit, δηλαδή ε, μας ε, ε, έθεσε πάλι σε επαγρύπνηση, ε, χτύπησε το κουδούνι του συναγερμού, οπότε δεν μπορούμε να λέμε ότι απλώς και μόνο επιτύχαμε το στόχο μας ε, και ε, επικρατεί η ειρήνη στην Ευρώπη. Θα πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και είδαμε πώς ψήφισαν οι νέοι στο πλαίσιο του Brexit και μάλιστα είχαμε και τη συντριπτική πλειοψηφία των των, των νέων. Και βέβαια εμείς είχαμε ταχθεί υπέρ του ακόμα και 16χρονοι να μπορούν να ψηφίζουν γιατί αυτό που συνέβη στο Brexit είναι οι μεγαλύτερε ηλικία γενιέ να αποφασίσουν για το μέλλον των νεότερων γενιών και τώρα οι νέε γενιέ θα πρέπει να δουν τι μπορούν να κάνουν για να ε, ζήσουν με το Brexit. Άρα λοιπόν ε, πραγματικά είναι πολύ ενεργή σε σχέση με τα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και θέλουν να έχουν λόγους στο πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ενότητας των υπολείπων έως 7 κρατών μελών, νομίζω πως σχετίζεται με αυτό που είπα μόλις τώρα, ότι δηλαδή θεωρούνταν ως κάτι το δεδομένο Ευρωπαϊκή υπολειπων ως οπότε βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα σοκ. Δεν αναμενόταν δηλαδή από κανέναν όλο αυτό. Και εγώ όταν άκουσα ότι θα γίνει ένα δημοψήφισμα, ήμουν σίγουρο ότι δεν θα χώρα και τελικά τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη ε, διαπίστωσαν ότι πράγματι αξίζει τον κόπο να διατηρηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, περνώντας στο τελευταίο ερώτημα που τέθηκε ως προς το τι ακριβώς σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση για μας, για τους νέους. Ε, νομίζω πως σε σχέση με αυτό είναι σημαντικό οι νέοι μα να νιώθουν εντό εισαγωγικών την Ευρωπαϊκή Ένωση καθημερινά. Για παράδειγμα, η δυνατότητα να μπορούμε να ταξιδεύουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο με την ε, ταυτότητά μα, το δελτίο ταυτότητα. Η δυνατότητα του να μπορούμε να ε, σπουδάζουμε, να εργαζόμαστε όπου θέλουμε, να αγαπάμε όποιον θέλουμε, να ε, παντρευόμαστε όπου θέλουμε. Οπότε είδαμε με, τους, ε, με το Brexit ε, το πώς οι νέοι άρχισαν να κάνουν μια επαναξιολόγηση των δικαιωμάτων τους, δηλαδή τι ακριβώς θα χάσουν με τη μορφή δικαιωμάτων. Χρειάστηκε λοιπόν να αξιολογήσουν, να ξαναδούν ποια είναι τα δικαιώματα των οποίων χαίρουν ε, και θέλουν να αγωνιστούν για αυτήν. Άρα λοιπόν δεν θεωρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, κάτι δεδομένο. Αντιλαμβανόμαστε το τι προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συχνά οι νέοι δεν έχουν ακριβώς τη δυνατότητα ε, και τις υποστηρικτικές δομές για να προσέλθουν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δουν τι ακριβώς ε, κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς. Αλλά παρότι ήδη κάνει κάποια πράγματα μπορεί ακόμα να καταδείξει ακόμα περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση το τι κάνει και μπορεί να αναλάβει και ένα πιο ηγετικό ρόλο και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη ως προς το τι μπορούν να επιτύχουν και πού βρίσκεται η περισσότερη προστιθέμενη αξία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, υπάρχουν κάποια ζητήματα ε, τα οποία για παράδειγμα είναι ασφάλεια τροφίμων ή άλλα ε, ζητήματα τυποποίηση ε, τα οποία εφαρμόζουμε, τα οποία δεν τα παρατηρούμε μέσα στην καθημερινότητα, τα οποία όμω τα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν λοιπόν ένα σωρό τέτοιοι λόγοι. Α συνεχίσουμε όμω τώρα Ας περάσουμε στη δεύτερη παρουσίαση με τον τίτλο Ευρωπαϊκή Ένωση, Δημοκρατία και Συμμετοχή. Ε, εν ώψη των επικίνδυνων ευρωεκλογών. Και έχω τον κύριο Νάζη εδώ ε, μαζί μας. Ε, και δεν έχουμε ουγγρικά σήμερα, αλλά ούτε ολλανδικά σήμερα. Γερμανία, το οποίο είναι κάπως ε, περίεργο. Βλέπω όμω στην Ολλανδική καμπίνα άδεια, οπότε ε, μπορείτε να μιλήσετε αγγλικά ή δεν ξέρω κάποια άλλη γλώσσα. Έχουμε ισπανικά, πορτογαλικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών εκλογικών νόμων. Είναι πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές εκλογές ε, για ε, τη δημοκρατία μας γιατί νομοποιούν το σύστημα διακυβέρνησης και διασφαλίζουν την ελευθερία στην Ήπειρό μας. Όμως, μόλις 42% ψήφισαν στις εκλογές του 2014 και αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και δεν λειτουργεί καλά στην δημοκρατία μας. Δεν έχουμε λοιπόν ευρωπαϊκή δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Έχουμε 28 διαφορετικά, διαφορετικές δημοκρατίες που ε, συναντιούνται κάθε πέντε χρόνια. Είναι σαφές αυτό όταν βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι δεν ψηφίζουν την ίδια ημέρη την ίδια μέρα. Υπάρχει ε, διαφορετικό εκλογικό όριο σε κάθε κράτος μέλος και δεν έχουμε καν την ίδια ηλικία μετά την οποία μπορεί κανείς να ψηφίζει. Ε, οι νέοι δεν εμπλέκονται στην πολιτική σκηνή γιατί σπάνια βλέπουν ε, κάποιον δικό τους ή της ηλικία τους να εκλέγεται. Όλες αυτές οι διαφορές καθιστούν πιο δυσνόητη την κατάσταση για τον απλό πολίτη και συχνά όταν κάποιος δεν κατανοεί κάτι, το αποφεύγει κιόλα. Γι' αυτό και είναι τόσο χαμηλή ε, η συμμετοχή σε εκλογέ. Γι' αυτό εσείς ε, πρέπει να αναλάβετε αυτό το έργο της μεταρρύθμιση. Οι ε, λίστες ε, δεν πέτυχαν, όμως πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια ε, του εκλογικού καταλόγου, να έχουμε μία ενιαία μέρα και ηλικία αλλά μπορούμε να πάμε ακόμα παραπέρα. Σε ό,τι αφορά τι ευρωπαϊκέ εκλογέ, λοιπόν, πρέπει να αφήσουμε κατά μέρο ε, τα εθνικά σύνορα και να έχουμε διασυνοριακέ εκλογικέ περιφέρειε. Φανταστείτε λοιπόν περιπτώσεις όπου μπορούμε να έχουμε ε, τους εκλογείς και από τις ε, δύο πλευρές των συνόρων που να συμμετέχουν σε εκλογές για την ίδια εκλογική περιφέρεια. Αυτό θα δημιουργήσει και ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης, ε, θα, έχει, θα δώσει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα και θα ενισχύσει τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές. Δώστε μας λοιπόν ε, τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ψηφίσουμε με έναν ευρωπαϊκό τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Για το Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, Πολιτικής Εκπαίδευσης, που βέβαια το center, το κέντρο, το γράφεται με την αμερικανική προφορά, αλλά ας πούμε ότι μιλάτε για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να απευθύνω το λόγο στην ε, Επιτροπή σας με προσκαλέσατε σήμερα για να σας μιλήσω για αυτή την πρόταση για, την Ευρωπαϊκή, για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής Εκπαίδευσης. Αλλά δεν θα μιλήσω γι' αυτό σήμερα, γιατί υπάρχουν πιο πιεστικά ζητήματα. Ήθελα σήμερα να σας μιλήσω στην ουγγρική γλώσσα, τη μητρική μου. Ε, φυσικά δεν φταίνε οι διοργανωτές που έκαναν ό,τι μπορούν για να υπάρχει διερμηνία. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ να το πράξω εξαιτία έλλειψη πόρων. Πώς λοιπόν μπορούμε να ε, αναμένουμε από άλλους Ευρωπαίους πολίτες που δεν μιλούν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά να συμμετέχουν ε, στις διαβουλεύσεις και τις πολιτικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν αποκλείονται από γλωσσική άποψη. Γι' αυτό θα ήθελα να σας μιλήσω για μια διαφορετική ε, πρόταση που είναι ένα κέντρο γλωσσικής πολυμορφίας και θα διασφαλίζει ακριβώς ε, την πολυγλωσία στην Ευρώπη. Ε, κάτι που συνάδει και με την αρχή της επικουρικότητας ε, θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση, υποδομές και υλικά προς τους νέους, προς τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών και φορείς που προάγουν την πολυγλωσία όπως τα τα μεταπτυχιακά και οι σχολές διερμηνίας, γιατί όλες οι γλώσσες έχουν ε, τα δικά τους προτερήματα και τη δική τους ομορφιά. Εγώ θέλω να ζω σε μια Ευρώπη που θα είναι αυτό που είναι, ε, ενωμένη στην πολυμορφία της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να θέσω ορισμένα ερωτήματα. Το κύριο Χοφμάιστερ πρώτα. Εκλέγονται ορισμένοι νέοι Συμφωνούμε όλοι ότι οποιοδήποτε 130 είναι νέος. Δεν το είπατε, αλλά προτείνετε ποσόστοση. Όχι, εντάξει, συμφωνούμε. Εσύ, εσείς, πώς ε, προσδιορίζετε ακριβώς την προστιθεμένη αξία των ε, υποψηφίων κάτω των 30 ετών. Δεύτερον, για την εναρμόνιση. Οπότε, πού σταματάει η εναρμόνιση και πού ξεκινάει η υπερβολική συγκέντρωση. Και δεύτερον, πώς θα πετύχατε μια τέτοια εναρμόνιση όταν υπάρχει τέτοια διαφοροποίηση μεταξύ των ευρωπαϊκών ε, πληθυσμιακών κατηγοριών. Θα το κάνετε με το ζόρι? Θα είναι μια διαδικασία που θα περάσει σιγά σιγά, γιατί ξέρετε, μέχρι να περάσει η διαδικασία μπορεί και εσείς να μην είστε πια νέος. Και μετά, εντάξει, κύριε Νάγκη, είναι μεγάλη, μεγάλος ο πειρασμός να μιλήσω και εγώ γκρικά, αλλά θα το κάνω. Σας ευχαριστώ που μιλήσετε και σε τόσες διαφορετικές γλώσσες. Εγώ φυσικά και είμαι υπέρ της πολυγλωσσίας, είναι προφανές. Υπάρχουν δυσκολίες με όλα αυτά που έχω διαβάσει εγώ για την κοινωνική ψυχολογία, δείχνει ότι υπάρχει μία κύρια γλώσσα στον εγκέφαλό μας και μετά οι υπόλοιπε είναι επικουρικές. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη πολυμορφία και στην χρήση γλωσσών και στην εκμάθηση και την κατάρτιση. Νομίζω ότι δημιουργεί έτσι αυτή την ε, γλωσσική ε, ποικιλότητα. Πώς έχουμε την βιοπικιλότητα, κάπως έτσι. Γιατί κάθε γλώσσα έχει έναν δικό της τρόπο ερμηνείας μιας λέξης. Ε, υπάρχουν λέξεις που μπορούμε να τις πούμε μόνο στα αγγλικά, άλλες μόνο στα αγγλικά. Βέβαια και τα αγγλικά δεν είναι μια ενιαία γλώσσα, υπάρχουν τουλάχιστον έξι. Το να έχουμε λοιπόν ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Γλωσσικής ε, Πολυμορφίας ε, θα με έβρισκε σύμφωνο. Απλώς ε, μπορεί αυτό το έργο τελικά να μην οδηγούσε στην πολυμορφία, αλλά στο αντίθετο, γιατί θα υπήρχε μια επιβολή της ομοιομορφίας. Αλλά το αφήνω στον ερωτηματικό. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Έχω δύο σύντομα σχόλια, λέει ο πρωτα Πρώτα-πρώτα, σε σχέση με την πρόταση, την ιδέα το ότι στις ευρωεκλογέ θα υπάρξει ευκαιρία να ψηφίσουμε ε, ευρωβουλευτές ε, που να αντιστοιχούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχουμε αυτά δηλαδή τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια. Πρόκειται για πρόταση που την έχει απορρίψει το Κοινοβούλιο φέτος. Δυστυχώς. Και ο υποφαινόμενος και η πολιτική μου ομάδα, οι σοσιαλδημοκράτες, ήμασταν υπέρ αυτής της πρότασης και άλλες ομάδες. Όμως η πλειοψηφία θεώρησε ότι αυτή η ας την πούμε φεντεραλιστική πρόταση δεν είναι υλοποιήσιμη. Και θεωρώ ότι ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο υπερεθνικό και επικεφαλής να έχει ε, τον υποψήφιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επρόκειτο να δώσει έναν μανδύα ε, υπερεθνικό όσον αφορά τις ευρωεκλογέ. Δυστυχώς όμως δεν συγκεντρώθηκε απαραίτητη πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο. Το γιατί έγινε αυτό να στο πούν άλλοι. Το θέμα είναι πώς ε, μας βλέπετε εσείς. Συνεχίζετε να πιστεύετε ότι τα κόμματα και τα ψηφοδέλτια των κομμάτων είναι το μέσον ε, που θα οδηγήσει στο να εκφραστεί η πολιτική σας επιλογή. Για πέστε μας πώς το βλέπετε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πασκάλ Ντυρό. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πρόεδρο. Δεν συμφωνώ με το ότι οι γλώσσες θα πρέπει να έχουν κάποια ομοιογένεια και να υπάρχει μία λίγκουα φράγκα γιατί νομίζω ότι έτσι έχουμε εξίσωση προς τα κάτω. Τελικά χρησιμοποιούμε τα κάποια αγγλικά. Κάποια αγγλικά όμως τα οποία ε, είναι τέτοια που δεν μπορούμε να εκφράσουμε κάποια λεπτά ε, ε, κάποιες, λεπ, κάποιες σκέψεις πιο περίπλοκες άλλωστε υπάρχουν οι μεταφραστές και μπορούν να κάνουν τη μετάφραση οπότε τελικά πρόκειται για ένα ταλέντο που δεν το έχουν όλοι και δυστυχώς διαπιστώνω ότι πολιτική σημαίνει το να κάνει κανείς επιλογές και εμείς εδώ για λόγους ε, έχουμε όλο ένα και λιγότερη μετάφραση. Να, σήμερα έχω ένα τριμερή διάλογο. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για ένα νομοθέτη παρά ο τριμερής διάλογος γιατί εκεί έχουμε τα τρία θεσμικά όργανα, κοινοβούλιο, συμβούλιο κλπ. Οπότε ε, δεν πρόκειται να έχουμε διερμηνία, δεν θα υπάρχει ερμηνεία στην σημερινή συνεδρίαση. Ε, και εγώ αρνούμαι να κατέβω σε μια τέτοια συνεδρίαση που θα ληφθούν κάποιε αποφάσει για την νομοθεσία και εκεί δεν μπορώ να εκφραστώ στη γλώσσα μου. Με βάζουν να μιλήσω σε μια άλλη γλώσσα. Ναι, εντάξει, μιλώ αγγλικά, αλλά δεν μπορώ να, να μπω στι λεπτομέρειες και αυτό νομίζω ότι είναι μια ανομαλία και θα διαμαρτυρηθώ, βεβαίως δεν θα τους καίγεται καρφί ως συνήθως, και προς τον πρώτο κοινοβουλίο δεν είναι δυνατόν να έχουμε χωρίς διερμηνία τέτοιες συναντήσεις αυτά αφορμή αυτά που είπατε για τα αγγλικά γιατί πρόκειται για έναν πλούτο για όλες αυτές τις ε, γλώσσες που έχει η Ένωση όμως, όμως αυτός ο πλούτος σιγά σιγά σβήνει και οδηγούμεθα σε κάποια μέτρια αγγλικά που δεν μπορεί να δώσουν κάποιες αποχρώσεις κλπ. Αυτό ως παρένθεση Τώρα στην ερώτησή μου θα προχωρήσω. Δεν ήμουν εδώ από την αρχή της συνεδρίασης και συμπαθάτε με, αλλά μιλήσατε για ε, την νεολαία, για το ότι δεν συμμετέχει ουσιαστικά σε ευρωεκλογέ. Όσον αφορά την γαλλική νεολαία, ναι, είναι μικρή η συμμετοχή. Και έχουμε το εθνικό μέτωπο Δεν μιλάμε τώρα για το εθνικό μέτωπο θα μπορούσαμε να το επικρίνουμε, αλλά πέστε μας τι σας φέρνει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πού σας αγγίζει. Ε, τι θεωρείτε ότι σας φέρνει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα ερώτημα που ασχολεί κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να μιλήσω και εγώ γερμανικά, εφόσον όλοι μιλούν τη μητρική τους. Για να μην μιλάμε όλοι κακά αγγλικά. γιατί πράγματι η γλώσσα αποτελεί πολυμορφία, αποτελεί πολιτισμό και ε, μία από τις βαθικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς ε, το να γνωρίζουμε καλύτερα εξοικείωση δηλαδή με τις γλώσσες και τους πολιτισμούς των υπολείπων ε, κράτων μελών. Άρα λοιπόν και με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θα πρέπει να αποτελέσει μια βασική μας κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει να καταστήσουμε όλα ίδια, ας μην τυποποιήσουμε τα πάντα. Και από εκεί και μετά βέβαια τίθεται το ερώτημα του πώς μπορούμε να μεταφέρουμε από τις πρωτεύουσε στις ε, αγροτικές περιοχές, ε, στην Ήπεθρο, ε, τις διαδικασίες, τις πολιτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί παντού σε, στις χώρες μας έχουμε για παράδειγμα τις ίδιες μεγάλες αλυσίδες όπως το Lidl ή άλλα σούπερ μάρκετ μεγάλα ε, τα οποία υπάρχουν και στις αστικές περιοχές και στις αγροτικές περιοχές ε, γιατί δεν κάνουμε κάτι αντίστοιχο ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δηλαδή δεν επιτρέπουμε στους ανθρώπους σε όλες τις περιοχές να συναποφασίζουν σε ό,τι αφορά την οικονομική και την κοινωνική τους πραγματικότητα. Δηλαδή πρόκειται για μια για περισσότερη ένδυα, αν θέλετε. Δηλαδή, γινόμαστε πιο φτωχοί όταν δεν υπάρχει μια τέτοια συμμετοχή σε αυτή την πολιτική διαδικασία. Νομίζω πω θα πρέπει να το θέσουμε αυτό το ερώτημα στον εαυτό μα. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι το πώ ακριβώ ψηφίζουμε. Εγώ ε, και η δική μου πολιτική ομάδα είμαστε υπέρ αυτών των διεθνών ε, ληστών, δηλαδή υποψηφίων για τι εκλογέ. γιατί είναι σωστό αυτό που υπόθηκε, ότι δηλαδή όταν λαμβάνουν χώρα ευρωεκλογέ, αυτέ λαμβάνουν χώρα σε 28 ή τώρα 27 κράτη-μέλη ξεχωριστά σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή δεν τίθεται ε, επιτάπητο σε ένα ζήτημα ή γενικότερα ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντο. Ε, γίνονται ε, ουσιαστικά ένα είδο δεύτερων εκλογών θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ευρωεκλογέ όπου υπάρχει ακριβώς επιρροή και στο τι ακριβώς κάνουν για τα συμβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικότερα με, την, ε, με, την, ε, με τις εξουσίες που έχει σε ό,τι αφορά τη συνομοθεσία. Γι' αυτό το λόγο νομίζω πως ε, θα πρέπει πράγματι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθούμε εντατικά με την αναδιατύπωση και την αναθεώρηση των εκλογικών κωδίκων, γιατί σε διαφορετική περίπτωση διαιωνίζουμε ουσιαστικά το πρόβλημα και τα κενά που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Ο λόγος και πάλι στον κύριο Χοφμάιστερ. Ευχαριστώ πολύ. Η προστιθέμενη αξία των νέων κάτω των 30 ετών. Δεν είναι θέμα ηλικίας, να σας πω πρώτα. Το θέμα είναι αν κάποιος ε, ξέρει τι κάνει. Αλλά τουλάχιστον για τη γενιά μου, το να βλέπουμε νέους ανθρώπους να εκλέγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει η αίσθηση ότι η Βρυξέλλες και γενικά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι κάτι το απόμακρο και ότι οι μεγαλύτερη σε ηλικία είναι εκείνοι που αποφασίζουν για εμάς τους νέους. Αλλά παρότι μπορεί να έχουμε κάποιους εκπροσώπους, δεν θεωρούμε ότι ακούγεται πραγματικά η φωνή μας εδώ. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό, δεν θέλω να γενικεύσω, αλλά το να έχουμε περισσότερους νέους ε, στην πολιτική θα ενθάρρυνα ακόμα περισσότερους να συμμετάσχουν. Το δεύτερο ερώτημά σας αφορούσε την εναρμόνιση και την ε, υπερβολική συγκέντρωση, η επιβολή. Ξέρετε ότι η εναρμόνιση συνήθως έχει θετικό αντίκτυπο. Τώρα εδώ πρέπει να δούμε πώς θέλουμε να εκλέγονται αυτοί οι άνθρωποι. Σε εθνικό επίπεδο, πολίτες της Βουλγαρίας, ε, της Γερμανίας της Ελλάδας ή ως Ευρωπαίοι. Εγώ θεωρώ ότι το δεύτερο πρέπει να γίνει. Να εκλέγεται κανείς ως Ευρωπαίος πολίτης. Και το να έχουμε 27-28 διαφορετικά εκλογικά συστήματα ουσιαστικά οδηγεί το να μην είναι ακριβώς ίσοι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ένας Γερμανός πολίτης μου πηγαίνει στην Κροατία και είναι εκεί κατά τη διάρκεια των εκλογών. Μπορεί να ψηφίσει διαλληλογραφία. Αν ένα Σλοβάκο πάει στο ίδιο ξενοδοχείο την ίδια ημέρα, δεν μπορεί να ψηφίσει γιατί ο Εθνικός Εκλογικός Κώδικας δεν επιτρέπει την ε, ψήφο διαλλογραφίας. Δεν υπάρχει λοιπόν ισότητα στα δικαιώματα των ε, εκλογέων. Δεν θέλουμε λοιπόν να επιβάλλουμε κάτι, απλώς θέλουμε να, είμαστε, να ασφαλίσουμε πραγματική ισότητα. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε για τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια. Θα μπορούσαν ε, πραγματικά να υπάρξουν. Τώρα για τα εκλογικά κόμματα που αναφέρατε. Και τις πολιτικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ο καθένας ψηφίζει το κόμμα του στη χώρα του. δεν έχουμε ευρωπαϊκά κόμματα που να έχουν, τις, να, είναι, να έχουν την ίδια μορφή και τις ίδιες αξίες όλα τα κρατη Είναι θέμα χρόνου βέβαια πιστεύω. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και για ιστορικούς λόγους ε, καθυστερεί αυτή η διαδικασία. Θα μπορούσαμε όμως να φανταστούμε κάτι τέτοιο στο μέλλον. καλύτερη εναρμόνιση και συγκερασμό των κομμάτων. Κύριε Ντιουγάν, τι μα συνδέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Είμαι Βουλγάρος, είμαι Γερμανός, ε, μιλάω όμως και τις δύο γλώσσες. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα αποτελεί τμήμα της ταυτότητάς μου. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ο κανόνας, οι περισσότεροι έχουν μία υπηκότητα και μια ταυτότητα. Όμως αυτό δεν αλλάζει. Παράλληλα όμως η γενιά μου είναι η γενιά του Εράσμους που παίρνει το ε, τρένο και μέσα σε τέσσερις ώρες βρίσκεται σε, σε άλλη χώρα, σε άλλο κράτος μέλος, ε, χωρίς ε, να περάσει από έλεγχο στα σύνορα. Και αυτό η γενιά μας το ξέρει, το αναγνωρίζει. Αυτό ακριβώς μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πράγματι Ευρωπαίοι. Και κύριε Σόλτς, να απαντήσω σε εσάς και στα γερμανικά. Συμμερίζομαι την ε, τοποθέτησή σας ε, στο ακέραιο και νομίζω πως ε, πραγματικά θα ήταν πολύ χρήσιμο το να έχουμε τέτοιου είδους διεθνείς εκλογικές λίστες γιατί και εγώ θεωρώ πως οι ε, επόμενες ευρωεκλογές ε, θα επιφέρουν πολλές αλλαγές, ε, γιατί δεν πρόκειται μόνο για το Brexit. Βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία όπου υπάρχουν πολλά νέα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει και η νεολαία του σήμερα. Οπότε πραγματικά συμφωνώ τα μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου αρχικά να επενέσω τους, ε, και, τους δερμηνείς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και νομίζω ότι η πρότασή μου για ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Γλωσσικής Πολυμορφίας μπορεί να μην είναι η μοναδική λύση, να είναι μία όμως από τις λύσεις και να μας δώσει τους πόρους που χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτή την εξαιρετικά πολύτιμη δουλειά που είναι απαραίτητη σε καθημερινή βάση για να απαντήσω στο ερώτημά σας, με ευρωβουλευτή. Το ιδανικό θα ήταν ένα Φιλανδό, ένα Σουηδό, ένα τσέχο, ένα Εστονό ή λιθουανό πολίτη που αυτή τη στιγμή ε, βλέπουν αυτή τη συζήτηση στο διαδίκτυο να είναι σε θέση να ακούσουν τα όσα λέμε και να σχολιάσουν στο διαδίκτυο ή να έρθουν και εδώ αυτοπροσώπους και να μιλήσουν στη γλώσσα του. Γιατί όπω λέτε πολλά χάνονται στη μετάφραση. Ε, πολύ, μεγάλη αξία, πολλέ μνήες, πολλές ε, αποχρώσεις. Με ρωτήσατε τι σημαίνει για μένα να είμαι Ευρωπαίος. Ο Σούγκρος για μένα αυτό είναι μία διασφάλιση ότι στον 21ο αιώνα θα διατηρήσουμε ε, το βιωτικό μας επίπεδο, τον τρόπο ζωής μας, να διατηρήσουμε την γλώσσα μας που τη μιλούμε εδώ και εκατοντάδες χρόνια και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για έναν πολίτη που πληρώνει φόρους και εκπροσωπείται εδώ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μιλήσει, και να ακούσει ε, στη γλώσσα του και να είναι σε θέση να συνομιλήσει με το Κοινοβούλιο. Από εκεί πρέπει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι, γιατί στον 21ο αιώνα είναι πολύ πιο εύκολο πλέον να ε, συμμετέχουμε σε αυτή τη δικασία. Ένας νέος μπορεί ε, μέσω του κινητού του να δημιουργήσει μια αίτηση Ευρωπαίων πολιτών, μια πρωτοβουλία, να συμπληρώσει ένα έγγραφο της διαβούλευση, ε, της Κεντρικής τράπεζα, για παράδειγμα. Όλα αυτά μπορούν να τα βρουν στα τάμπλετ, στα κινητά και στα λάπτοπ. Σύμφωνα όμως με το Ευρωβαρόμετρο 89,2, το 34% των ε, πολιτών μας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν το 34% θεωρεί ότι ο κόσμος δεν ψηφίζει γιατί δεν κατανοεί πραγματικά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει επειδή οι Ούγγροι συμπατριώτες μου που μπορεί να μας παρακολουθούν δεν θα καταλάβουν τι γίνεται εδώ σήμερα αν δεν είχαν την ευκαιρία να μάθουν αγγλικά. Γι' αυτό και ελπίζω κάποια στιγμή να είμαι σε θέση να σας επευθύνω το λόγο στη μητρική μου γλώσσα και αυτή η δυνατότητα να, να δίνεται σε ολόκληρο το Ευρωκοινοβουλίο κοινοβούλιο που εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Να προσθέσω κάτι για την έλλειψη Ουγγρικών. Στην προηγούμενη θητεία είχαμε Ουγγρικά, γιατί είχαμε και τρεις Ούγγρους βουλευτές. Σε αυτή τη θητεία είμαι ο μοναδικός Ούγγρος ευρωβουλευτής και τα αγγλικά μου πέντε λες και άσχημα, γι' αυτό αποφασίσαμε να μην έχουμε Ουγγρικά. Υπάρχουν λοιπόν ειδικέ ε, περιστάσεις, δεν χρειάζεται να, το, ε, να κατηγορούμε την Επιτροπή. Ο αντιπρόεδρος είναι εδώ και μπορείτε να μιλήσετε και την γλώσσα σας. Τα δανεικά. Εντάξει, θα συνεχίσω. Η τρίτη θεματική κατηγορία διατήρηση και βελτίωση ενός δίκαιου και διαφανούς ευρωπαϊκού χώρου συζήτησης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες. Παρακαλώ, διατηρήστε και κρατήστε το όριο των ε, δύο λεπτών. Παρακαλώ, έχετε λόγο. Η δεύτερη ιδέα λοιπόν που προτείνω είναι να γίνει με αναθεώρηση του ε, συστήματος υποβολής ε, ε, αναφορών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πως ε, το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα υποβολή αναφορών αποτελεί μια καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εισήχθη για πρώτη φορά στο Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο το 1999 και έκτοτε υπάρχει στην Κάτω Βούλη τη Γερμανία, του Ηνωμένου Βασιλείου και τώρα και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και προκειμένου λοιπόν τώρα να βελτιώσουμε αυτό το μοναδικό εργαλείο συμμετοχή δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ θα ήθελα να προτείνω τρει μεταρρυθμίσεις, αν θέλετε, βασιζόμενες στις εμπειρίες των κρατών μελών. Καταρχήν, α δημιουργήσουμε ένα online forum. Ε, δηλαδή, στην Γερμανική Κάτω Βουλή, η ε, πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τα πλέον εκτήματα και τα μειονεκτήματα τέτοιου είδου ε, ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων αναφορών. Ένα τέτοιο λοιπόν φόρουμ θα επέτρεπε στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν μια ποιοτικότερη συζήτηση, ένα διάλογο μεταξύ τους σε ό,τι αφορά ε, τις αρετές αλλά και τα ανεδικά στοιχεία μια αναφορά. Επίση, α μειώσουμε το σχετικό κατόφλη σε ό,τι αφορά μία αναφορά. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, εάν συγκεντρώσει 100.000 υπογραφέ μία αναφορά, θα πρέπει να εξεταστεί από την κάτω βουλή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ήθελα λοιπόν ε, το ίδιο κατόφλι να ισχύσει και για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, για το δικό μα κοινοβούλιο, έτσι ώστε να δίνουμε μία υποχρεωτική απάντηση στις, σε αυτά τα ερωτήματα των πολιτών μα. Και επίση, τρίτη μου πρόταση είναι να έχουμε περισσότερε ακροάσει με βάση δηλαδή ε, το Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο ε, ε, και το παράδειγμά του γίνεται πρόσκληση των πολιτών σε σχέση με τις αναφορές. Αλλά εγώ θα ήθελα να προτείνω να έχουν τη δυνατότητα εν λόγω πολίτες να προσέρχονται εδώ στο κοινοβούλιο και να γίνεται μια ακρόασή τους τόσο σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω πως θα μπορούσατε να πραγματικά υποστηρίξετε ε, ένα τέτοιο project ώστε να, υπάρξει, να ξεκινήσει με εποχή μεταρρυθμίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, να μας ε, αναφέρετε κι εσείς ε, τώρα την πρότασή σας σε ό,τι αφορά την τηλεοπτική συζήτηση, τον πολιτικό διάλογο. Ναι, αυτό που προτείνουμε είναι ακριβώ προκειμένου να βελτιωθεί ο διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε ε, στο πλαίσιο και τη εκπαιδευτική ανάληψη ε, τη Προεδρία κάθε 6 μήνε σε μια τέτοια τηλεοπτική συζήτηση. Γιατί νομίζω πω ε, βασικέ αρχέ εδώ είναι η δημοκρατία και με βάση ακριβώ και την πολυγλωσία την οποία προωθούμε είναι πιο εύκολο από ποτέ. Έχουμε δηλαδή κάνει κάποιε προσπάθειε και με το Άρτε, για παράδειγμα, το τηλεοπτικό κανάλι ή το Euronews, αλλά με πιο περιορισμένη επιτυχία. Ας λοιπόν κάνουμε κάτι τέτοιο τώρα, μια αντίστοιχη προσπάθεια με ένα πιο ενδιαφέρον ζήτημα. Καθώ και η περιτροπή ανάληψη τη Προεδρίας είναι κάτι το μοναδικό, γιατί δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί δηλαδή δεν έχουμε μια τέτοια τηλεοπτικά αναμεταδιδόμενη συζήτηση κάθε έξι μήνε όπου οι διάφοροι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων ε, και των κρατομελών συζητούν τι ε, ε, προτεραιότητε τη επόμενη προεδρία. Αυτό λοιπόν, αυτή η τηλεοπτική συζήτηση θα γίνεται, θα αναμεταδίδεται live, ζωντανά δηλαδή, μέσω web stream streaming και έτσι θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν αλλά και βέβαια και, στις, ε, και στον τύπο. Με αυτόν τον τρόπο, ε, με αυτή την αναμετάδοση νομίζουμε ότι θα υπάρξει συμβολή στον γενικότερο πολιτικό διάλογο, στον πολιτικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε πως ε, τα, η, κάθε Προεδρία καλείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της για κάθε έξι μήνες, αλλά φανταστείτε να έχουμε μια τηλεοπτική συζήτηση με υψηλό βαθμα στελέχη, χύνοντες πολιτικούς, όπου που θα γίνεται μια συζήτηση μπροστά στι κάμερε σε σχέση με τα σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα. Νομίζω πω μια τέτοια συζήτηση θα μπορούσε να συμβάλλει σε περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη ευαισθητοποίηση ε, και περισσότερη συμμετοχή εμπλοκή στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Νομίζω πω κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου αυτή να λειτουργήσει. Α δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία στου ε, πολίτε μα να αντιληφθούν τι ακριβώ συμβαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε. Ερωτήσεις από τους συναδέλφους ο κύριος Χάρηγη πολύ σύντομα. Πρώτα πρώτα ευχαριστούμε για τις ε, προτάσεις σας. Μερικές ε, από αυτές πολύ ενδιαφέρουσες και θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη για τη δουλειά μας στο μέλλον. Ήδη κάποια που αναφέρετε τα κάνουμε. Έχουμε την Επιτροπή Αναφορών εδώ στο Κοινοβούλιο που είναι αποδέκτης ε, κάθε μήνα δεκάδες φορείς από όλη την Ευρώπη που έρχονται και λένε το πρόβλημά τους άμεσα. Εδώ στο Κοινοβούλιο γίνεται αυτό πολύ συχνά και υπάρχει αυτή η συζήτηση που, θα γίνει, που έγινε μάλλον το Σεπτέμβριο για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και νομίζω ότι πρόκειται να υπάρξουν και άλλες ε, συζητήσεις και διάλογος μεταξύ των επικεφαλής υποψηφίων για τις εκλογές και η ιδέα αυτή του να χρησιμοποιείται η τηλεόραση για να έρχεται πιο κοντά ο κόσμος στο κοινοβούλιο αυτό ε, είναι κάτι δεδομένο ως ιδέα και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία που έχουμε. Συμφωνούμε 100% με ό,τι είπατε. Thank Απλώς να σας πω ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία για τα νέα μέσα ε, για τους ε, Ευρωπαίους τα ξέρει ο κύριος Σέφλιν ότι αυτά ήδη βρίσκονται εδώ ε, από τη στιγμή της Λισαβόνας και μετά το έχουμε κάνει και οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτές τις πρωτοβουλίες των πολιτών και το, το χειρότερο είναι το ότι θα πρέπει κανείς να μπορεί να έρχεται σε επαφή με τους έρετους άρχοντες αλλά το χειρότερο είναι μετά από αυτό να μην κάνουν τίποτα αυτοί να, γιατί αξίζει η πρωτοβουλία των πολιτών. Τώρα για τους καντιντάτεν, αυτούς τους επικεφαλής, τους κορυφαίους υποψηφίους, ε, είπαμε για να γίνει κάποιο είδου ε, debate, να μεταδοθεί στις τηλεοράσεις σε όλες τις χώρες. Το θέμα είναι πόσοι παρακολουθούν αυτά τα debate. Γιατί αν υπάρχει απογοήτευση, ε, δεν κάνει κανείς τίποτα με τα μέσα επικοινωνίας. Οπότε αυτό θα πρέπει η γενιά σας να αντιμετωπίσει. Το πώς θα, θα ξυπνήσει το ενδιαφέρον. Ε, η αίσθηση του, να είναι κανείς Ευρωπαίος. Ιταλός, Γάλλος. Ε, βέβαια, ε, κανείς ανήκει στην Ευρώπη, είναι Ευρωπαίος, αλλά ε, υπάρχει και αδιαφορία. Αυτά λέω στα παιδιά μου που έχουν την ηλικία σας. Το μέσο αυτό θα δούμε για το πώς θα, έρθει κοντά σε αυτή την ιδέα της, στον προορισμό αυτών η νεολαία. Γιατί οι τεχνοκράτες δίνουν τα μέσα, αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα μέσα. Οι δάλλοντες δεν ωφελούν. Επομένως, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα στην ε, Ευρώπη. Αυτό είναι το έλλειμμα. Ε, ψυχή και καρδιά λείπουν. Δεν λείπουν τα μέσα, τα εργαλεία. Άρα, ακριβώς αυτό θα πρέπει να υπάρχει. Ο πόθος, η επιθυμία για τον κοινό προορισμό, το κοινό μέλλον. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό στα πλαίσια της λειτουργίας της Ένωσης. αυτό που αποτύχαμε ε, να, το, να το δώσουμε, να το μεταλαμβαδεύσουμε στους ε, Βρετανούς, στο κοινό μέλλον. Σόφλιν. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω κάποιες σκέψεις μου. Ο ρόλος των ΜΜΕ. Δυστυχώς, τα μέσα Συνήθω ασχολούνται με την διμερή ούτως ποινή πολιτική, όχι την ευρωπαϊκή πολιτική. για τις σχέσεις Γαλλίας-Γερμανίας ας πούμε. Πότε ακούστηκε η Πορτογαλία γιατί ποτέ. Άρα, εσείς που ασχολείστε με την πολιτική στα κράτη-μέλη σας δεν έχετε την ευκαιρία να δείτε τι γίνεται εδώ στην Ευρώπη. Είναι και εγώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι. Δεν, δεν, δεν το κατάφερα. Αυτό θα πρέπει να υπάρξει για να προοδεύσουμε σε σχέση με το στόχο μας. Τώρα, όσον αφορά την πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ασυνείδηστο αυτό το Κοινοβούλιο. Πάντως, αρμοδιότητα της νομοθετικής πρωτοβουλίας την έχει η Επιτροπή και όχι το Κοινοβούλιο. Άρα εδώ διαφέρουμε από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Βέβαια, έχουμε την πρωτοβουλία των πολιτών που μας είπε ο Πασκάλ Τυρό. Έχω αναλάβει μια σχετική έκθεση, τώρα βρίσκομαι στην τελική ευθεία. Λειτουργεί αυτό σε Φιλανδία και Λετωνία, οπότε πολλοί πολίτες μπορούν να υπογράψουν ε, αυτή την πρωτοβουλία. Οπότε τα κοινοβούλια υποχρεούνται να τους ε, ακούσουν. Και αποφασίζουν να γίνεται ψηφορία γι' αυτό. Οπότε, να, ποιο είναι το θέμα με το κοινοβούλιο. Το ότι η Επιτροπή έχει την πρωτοβουλία και από εκεί ξεκινάνε όλα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. ε, κύριος μετά και τώρα ο κύριος Νάγκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας, τα καλά σας λόγια και ήθελα να σας ε, πω κάποια προσωπική εμπειρία στην γνωστή εκδήλωση στην Ολομέλεια που έγινε είπα ότι Έχουμε νέους από την Ευρώπη, γεμάτη η αίθουσα και ρώτησα πόσοι από εσάς έχετε ε, υπογράψει μία ε, αναφορά λιγότερο από πέντε σήκωσαν το χέρι τους ε, ενώ όλοι είχαν τα μέσα τα τεχνικά για να το κάνουν αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία του 21ου αιώνα, θα πρέπει να βελτιώσουμε το εργαλείο αυτό να είναι ε, πιο ελκυστικό, να είναι πιο προσβάσιμο και έτσι και οι νέοι θα έχουν κίνητρο να ασχοληθούν και στο Μερο Βασίλειο βάλανε ένα κατόφλι 10.000 ε, υπογραφές για να δράσει η, η κυβέρνηση ή για κάποια αναφορά, για κάποια ακρόαση, 10.000 υπογραφές και ε, έγινε αυτό μέσω των ε, ε, κοινωνικών δικτύων. Πάρα πολύ καλό αυτό. Τώρα, όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος βουλευτής που ρώτησε, θα πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση μεταξύ της πρωτοβουλίας των πολιτών και των αναφορών που έρχονται εδώ. Και ο κύριος Σέπλιν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Υπάρχει εδώ διαφορά και Στη δική μας περίπτωση ο στόχος θα πρέπει να είναι οι να μπορούν να επισημάνουν, να αναδείξουν ένα θέμα και να επιδιώξουν την λύση του. Δεν αρκεί το να γίνονται επικρίσεις. Πρέπει να υπάρχει σωστή διάγνωση του προβλήματος, σημαντικό αυτό, αλλά θα πρέπει να έρθει και η λύση του προβλήματος. Και εσείς οι αιρετοί εκπρόσωποι αυτό μπορείτε να κάνετε και μία ένα από τα υπέρ τη ε, Επιτροπή Αναφόρων ότι μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί να αρχίσει να δίνεται η λύση. Αλλά πάντω είναι, είναι μια αφετηρία η αναφορά ε, για την ε, δημοκρατία στην Ευρώπη και θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Ε, πολύ σπουδαία παράδοση αυτή η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ όλου πάρα πολύ. Ο χρόνο μα τελείωσε. Α, συγγνώμη. Σα ξέχασα, κύριε ναι, μπορείτε να μακρηγορήσετε όσο θέλετε εντός δύο λεπτών. Ευχαριστώ. Και από το 2014 είχαμε ε, debate με τους speech and αλλά τι, αυτό αρκεί, όχι. Δεν νομίζω, γιατί εάν θέλετε να ελκύσετε, να, να, να στρατεύσετε ούτως του, τους νέους, δεν αρκεί αυτό να γίνεται κάθε πέντε χρόνια με τίποτα. Ε, τι, ίσως κάθε έξι μήνες που αλλάζει η συζήτηση, που αλλάζει συγγνώμη, η Προεδρία του Συμβουλίου. Αυτό να γίνεται, αυτό θα μπορούσε να ενδιαφέρει τον κόσμο ε, γιατί ε, έτσι, έτσι θα κερδίσετε ξανά την καρδιά των Ευρωπαίων επίσης. Σύντομα. Και για να είμαι πολύ σύντομο, ε, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως ε, αυτό εξαρτάται από τα εθνικά μέσα ενημέρωση Εσείς ε, ως Κοινοβούλιο και ω ε, Επιτροπή δεν μπορείτε να έχετε βέβαια κάποια επιρροή σε αυτό και αυτό είναι καλό βέβαια, αλλά μια τέτοια τηλεοπτική συζήτηση ανά έξι μήνες και η δυνατότητα το να το κάνουν τα μέσα ενημέρωση ουσιαστικά θα έδιναν μια περισσότερη δυνατότητα για ενδιαφέρον ε, στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα. Δηλαδή, αν κάθε έξι μήνες υπάρχει αυτή η πρόσκληση για μια τελευταία συζήτηση, τότε τα μέσα θα θεωρήσουν ότι αρχίζει πραγματικά κάτι και κινείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουν ήδη, απλώς δεν το βλέπουν. Οπότε το να έχουμε πραγματικά πολιτικούς υψηλού επίπεδου, ψηλόβαθμου, οι οποίοι συμμετέχουν σε τέτοιου είδου συζήτηση, πραγματικά θα προσέλκυε περισσότερο τα μέσα ενημέρωση και έτσι θα γινόταν περισσότερο πολιτικό διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο θεωρώ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο, ο Πρόεδρο. Ε, δεν είμαι τόσο πεπισμένο όσο εσεί ότι τα μέσα ενημέρωση αντιλαμβάνονται ε, την πραγματικότητα αυτή, δηλαδή την ε, πολιτική εξουσία ε, και την, την, το τι συμβαίνει σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας το λέω αυτό γιατί δούλεψα για νέα χρόνια ως δημοσιογράφος. δηλαδή συχνά τους είναι τελείως ξένη η ιδέα του, του υπάρχει ε, ε αμυγός ευρωπαϊκός χαρακτήρας σε ορισμένα ζητήματα. Αυτό νομίζω πως είναι το βασικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το να ε, μπορέσουμε να περάσουμε σε μια πραγματικά ευρωπαϊκό επίπεδο δημοκρατία και αποτελεί ε, καθήκον δικό σας της νέας γενιάς να αλλάξετε αυτή την κατάσταση. Πάντως σας ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες εδώ και την παρουσία σας ε, σήμερα εδώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις που έθεσαν και νομίζω πως είμαστε και μέσα στο χρονοδιάγραμμά μας. Ναι, έχουμε μόνο αργήσει πέντε λεπτά, πράγμα το οποίο είναι πολύ καλό με βάση τι συμβαίνει συνήθως στην Επιτροπή μας. So after this thorough discussion, μετά αυτήν την λεπτομερή συζήτηση, which of course had to be steered by one of the most experienced parliamentarians, uh, όπου είχαμε και μια σειρά από συναδέλφους που συμμετείχαν. Και αναλαμβάνω λοιπόν την Προεδρία τώρα για το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης που είναι η έκθεση από Μισελα Μασούρ που παρευρίσκεται εδώ στην αίθουσα. Σε ό,τι αφορά αυτό το σχέδιο έκθεση, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των συνδικών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία. Δίνω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή μα ε, για να παρουσιάσει αυτή την έκθεση και συνέχεια θα δώσουμε το λόγο σε όλου του συναδέλφου ε, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Παρακαλώ, κύριε Λαμασού. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριο Λαμασούρ αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση που έχω την τιμή να σας ε, παρουσιάσω σήμερα είναι το δεύτερο τμήμα του έργου που αναλάβαμε για να δούμε τις ε, νέες μορφές συνεργασίας των μελών. Ο Πασκαλντυρόν είχε ε, ολοκληρώσει το πρώτο τμήμα αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή να δούμε πώς έχει η κατάσταση σήμερα και τι δυνατότητες υπάρχουν στο μέλλον όσον αφορά την ενισχυμένη συνεργασία. Πολλούς μήνες δουλέψαμε με τους σκιώδεις ηγητές διοργάνωσε κάποιες ε, ακροάσεις η Επιτροπή μας ε, με όλα τα σμικά οργάνα και καλέσαμε υπαλλήλους είχαμε τον καθηγητή Βέσελς όσον αφορά την ε, εφαρμογή του θεσμού αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε και μελετή επιπτώσεων που την έκανε η υπηρεσία έρευνας του Κοινοβουλίου και έγινε και εντελεχής ανάλυση του θεσμού αυτού που υπάρχει και σε ομοσπονδιακά κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάναμε και δύο νημερωτικές αποστολές στην ε, Βέρνη της Ελβετίας για να μπορέσουμε να μελετήσουμε το τι γίνεται στα ελβετικά καντόνια. Τη συνεργασία έχουν τα καντόνια για όσα θέματα δεν είναι ομοσπονδιακής αρμοδιότητας. Και επίσης πήγα και στην Ουάσιγκτον για να δω πώς λειτουργεί εκεί το αντίστοιχο σύστημα στην ε, Αμερική για συνεργασία μεταξύ των Αμερικανικών πολιτιών. Δύο παρατηρήσεις ε, πάρα πολύ σημαντικές, πολιτικές όσον αφορά το πνεύμα και τον στόχο αυτής της έκθεσης. Δεν πρόκειται να αναφερθούν κάποια κράτη-μέλη συγκεκριμένα, ούτε, ούτε είναι θέμα πολιτικής ο στόχος. Δεν είναι να ενθαρρύνουμε τα κρατημέλη που επιθυμούν να έχουν μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων δύο κατηγοριών. Να έχουμε την Premier League από την πρώτη κατηγορία και την δεύτερη εθνική. Όχι, δεν πρόκειται περί τούτο. Επίσης, δεν είναι θέμα της Επιτροπής Δεγματικών Υποθέσεων να ε, αποφανθεί για το σε τι αρμοδιότητες, σε τι πολιτικές προσυδειάζει αυτή η ε, διαδικασία. Απλώ καθόμαστε και κάνουμε μια καταγραφή του τι ισχύει και το πώς αυτό το μέσο, το εργαλείο μπορεί να συμπληρώσει, να βελτιώσει, ε, να συγκεκριμενοποιήσει τα πράγματα να είναι πιο χρήσιμο στα πλαίσια των, ε, των συνθήκων για τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω για ποια, για, για ποιους, ποιες αρμοδιότητες δεν ξέρω, πως ώστε τέλος πάντων να είναι καλύτερη συνεργασία και ε, αυτό να γίνει ε, όχι με κυβερνητικές, διακυβερνητικές συμφωνίες όπως το δημοσιονομικό σύμφωνο εκτός συνθήκης δηλαδή για να φέρουμε κάτι πολύ σημαντικό, αλλά το πώς θα υπάρχει αυτή η συνεργασία μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι οι χώρες που θέλουν να συνεργαστούν περισσότερο για κάποια ε, συγκεκριμένες ε, κοινέ του αρμοδιότητες να μπορέσουν να το κάνουν ε, άπαξ και συγκεντρώνεται το 1 τρίτο των μελών και να γίνει αυτό μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτό το σύστημα ε, έτσι να οι αποφάσεις και να μπορούν ε, ε, στη ζήμωση αυτής της συνεργασίας να συμμετέχουν και άλλα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο και επί τη βάση των εμπειριών που ήδη έχουμε θα διαπιστώνουμε ότι για κάποια θέματα για τα οποία θα ήταν χρήσιμο, θα ήταν ευκταίο να υπάρχει τέτοια περισσότερη συνεργασία ας πούμε στο πνεύμα της ε, ΟΝΕ Πάντως υπάρχουν και άλλα θέματα για το οποίο δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Ας πούμε, εάν κάποιες ε, χώρες που βρέχονται από τη Βαλτική θέλουν να κάνουν κάποια ενισχυμένη συνεργασία, θα πρέπει να συγκεντρωθούν ε, εννέα ε, χώρες προς τούτο, αλλά θα μπορούσε να συμμετασχεί και η Μάλτα, η Πορτογαλία, χώρες της Μεσογείου. Οπότε, κάνουμε αυτές τις απαραίτητες ε, πολιτικές διευκρινήσεις. Πώς έχει τώρα η κατάσταση νομικά. Η συνθήκη της Λισαβόνας διευκολύνει την συνεργασία αυτή, τη διαδικασία αυτή. Αλλά δεν λέει πολλά όσον αφορά την ε, λειτουργία, την διαδικασία. Εδώ μπορούμε να έχουμε κάποια προσθέμενη αξία από δική μας πλευράς και έχουμε την ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, πρόταση της Κομισιόν, έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ενισχυμένη συνεργασία μπορεί να καλύπτει μια ε, συγκεκριμένη ρήτρα που λέγεται πασαρέλα, γέφυρα και πέραν αυτής της ειδικής πλειοψηφίας διευκρινίζεται ότι η οικονομική πτυχή του θέματος καλύπτει το, κάτι, κάποιες δαπάνες πέραν των δαπανών ε, λειτουργίας που αφορούν τα κράτη που συμμετέχουν άμεσα. Όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στις ε, ζυμώσεις συζητήσεις, αλλά μόνο τα μέλη αυτής της διαδικασίας μπορούν να αποφασίσουν. Μέχρι σήμερα είχαμε τέτοιες, ε, τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις όπου λήφθησαν αποφάσεις για διαφορετικά θέματα και από διαφορετικές χώρες. Είχαμε το νομοθέτημα για το διαζύγιο το οποίο το μόνο που εφαρμόστηκε πραγματικά. Επίσης έχουμε τους κανόνες σε σχέση με το γάμο και συναφή ζητήματα. Αυτό θα αρχίσει να ισχύει από την πρώτη πρώτη επόμενου έτους. Επίσης Ευρωπαϊκό Τύπο Ευρεσιτεχνίας χρειάζεται ε, κάποια συμπλήρωση όσον αφορά την δικαστική επίλυση των διαφόρων Και τελευταίο αλλά σημαντικό το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αυτό θα αρχίσει να λειτουργεί, να εφαρμόζεται από του χρόνου. Και επίσης έχουμε το θέμα της ε, ε, Επίσης και για την άμυνα έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις κάπως έτσι. Και παρουσιάζει ενδιαφέρον το εξή. Πολλά κράτη-μέλη τα οποία συμφωνούν σε αυτή τη συνεργασία είναι πάνω από τα 17 έως 26 έχουν, έχουν συμμετάσχει. Και αν ε, κάποια χώρα όπως το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία συμμετέχουν ε, σε όλες τις ε, ε, συνεργασίες διαπιστώνουμε ότι έχουν συμμετάσχει διαφορετικές χώρες και προέρχονται από παντού, από βορρά, νότο, ανατολή, δύση. Επίσης, διατηρούμε κάποιες ε, προτάσεις, και έτσι να αξιοποιήσουμε την ενισχυμένη συνεργασία. Είμαι πεπισμένος ότι για δύο κατηγορίες θεμάτων η συνεργασία των κρατών μελών βοηθά την ολοκλήρωση, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό θέμα που με απασχόλησε. Αυτό πάντως θα ενισχύσει την αίσθηση του ότι συμμετέχουμε σε ένα κοινό όραμα τους λαούς. Και πέραν τη έλλειψη ευελιξία, τη συνθήκη όσον αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων, μπορούμε να θεσπίσουμε κάποιες διαδικασίες που δίνουν ευελιξία και αφορούν κάποιες δράσεις, κάποιες ενέργειες και κάποια κράτη-μέλη. Είναι επομένω δύο κατηγορίες, όλο διαφορετικές κατηγορίε θεμάτων, πολύ σημαντικέ πολιτικά ασφάλεια, κάποια θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά. Δεν ε, το διευκρινίζω περισσότερο. Όμως μπορούν να καλυφθούν και άλλα θέματα που είναι πολύ πιο κοντά στον Ευρωπαίο. να σχετίζονται περισσότερο με τι εθνικέ αρμοδιότητες, ούτω ώστε να διευκολυνθεί η ζωή του πολίτη, οι δραστηριότητε των επιχειρήσεων, εναρμόνιση, ενοποίηση αυτών των αρμοδιοτήτων που θέλουν κάποιες χώρες. Μπορούν να επιλέξουν αυτή τη διαδικασία. Και επίσης εδώ δηλαδή, σε κάποια κράτη-μέλη όπως στην Γερμανία σε κάποια κράτη εκτός Ένωσης, είπα Ελβετία, τα καντόνια και οι Αμερικανικές πολιτείες έχουν θεσπίσει εδώ και έναν αιώνα ένα σύστημα συνεργασίας μεταξύ τους, μεταξύ ε, πολιτιών ή καντονίων. Και έτσι από κοινού ρυθμίζουν σε εκείνο το επίπεδο ότι χρειάζεται χωρίς αυτά τα θέματα να, ε, να πάνε στο κρατικό επίπεδο, στο κυβερνητικό επίπεδο. Ε, συμβόλαια, συμφωνίες λέγονται αυτά για τα καντόνια και στις ΕΠΑ είναι τα πολιτιακά σύμφωνα όπως τα λένε, state και πρόκειται για διαδικασίες που έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και υπάρχει και το νομικό ίδρυμα στη ΣΥΠΑ που έχει κωδικοποίησει τη διαδικασία οπότε το εμπορικό δίκαιο και ε, άλλα θέματα είναι πολιτικές αρμοδιότητες και όχι κρατικές. Σαράντα περίπου πολιτείες αποφάσισαν όχι απλώς να κάνουν εναρμόνιση αλλά να έχουν ακριβώς τον ίδιο νόμο, το ίδιο δίκαιο που να διέπει τις ε, πολιτείες. Και αυτά επί της αρχής με την ευλογία του Κογκρέσου που ψήφισε σχετικά. Και βέβαια ε, το το Δικαστήριο τον είπα, ασκεί εποπτεία. Οπότε θεωρώ ότι αυτές οι εμπειρίες μπορούν να μας εμπνεύσουν για το έργο μας, τα κράτη-μέλη εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι συγκρίσιμο το πνεύμα αυτών των ε, θεσμών Καναδάς και Αυστραλία επίσης ε, ενδιαφέρον και πήγαμε εκεί και οργανώσαμε κάποιες ε, ακροάσεις. Οπότε έχουμε εδώ αυτές τις έξι επιλογές, πολιτικές επιλογές που διέπουν την ε, λειτουργία αυτής της διαδικασίας, της ενισχυμένης συνεργασίας. Και έτσι διευκολύνεται η διαδικασία. Οπότε να βελτιωθεί ότι αποτελεί κακό κείμενο στην Ευρώπη ή εκτός Ευρώπης τυχόν και τελικά διαδικασία αυτή να έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Άρα αυτή είναι η πολιτική επιλογή, πώς θα γίνεται αυτή η διαδικασία, ποια θα είναι τα όργανα ε, που θα αποφασίζουν πρακτικά οι υπουργοί με αυτή την ειδική πλειοψηφία. Ποιο οργανώνει την ε, ε, γραμματεία, τι θα, θα είναι ad hoc, θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δεν είναι Επιτροπή, τι ρόλο θα πρέπει να παίζει υπέρ των κρατών μελών κατά την διαδικασία αυτή. Είναι και το θέμα της οικονομικής κάλυψης. Χρήσιμο το τι έγινε στην περίπτωση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, τι είδους κοινοβουλευτικός έλεγχος θα υπάρχει. Θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο ε, θα ασκεί κάποια αρμοδιότητα, όλο το Κοινοβούλιο, κάποια επιτροπή συγκεκριμένη του Κοινοβουλίου, ε, ανάλογα με το θέμα της συνεργασίας και όλοι να συμμετέχουν ε, στις συζητήσεις, επαφές, αλλά τελικά στην, αν θα συμμετέχουν όλοι ή όχι στην ψηφοφορία αν θα συνεργάζεται αυτός ο ρόλος όπως με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο του Ευρωκοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια και βέβαια να δούμε πώς θα γίνεται η δικαστική επίλυση των διαφορών. Ε, βέβαια, τελικά είναι, αποφαίνεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε και κάποιο είδους διαμεσολάβησης, ακριβώς όπως κάναμε και με το ε, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Ε, επίσης ποια είναι τα υπέρ και τα κατά αυτών των επιλογών και πόσο υλοποιήσιμες είναι αυτές οι επιλογές, αυτές οι λύσεις και ο στόχος είναι το πώς θα διευκολύνουμε τα κρατη που θα θελήσουν να προσφύγουν σε αυτή τη διαδικασία για κάποια θέματα. Επίσης, πολύ σημαντική πρόταση γίνεται στο ότι η Επιτροπή και το βούλιο ενδιαφέρονται ιδιαίτερος και, και οργανώνονται ούτως ώστε να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία όταν ξεκινάει. Όπως, ό, όποιος και να το ξεκινάει, εσύ το, ξεκινάει τη διαδικασία τα κράτη-μέλη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ενδιαφέρονται, να ασχολούνται με το θέμα Κοινοβούλιο και Επιτροπή. Κάτι που δεν ισχύει μέχρι τώρα. Μα και το ίδιο το Συμβούλιο επίσης τώρα δεν συμμετέχει τόσο Προεδρία Υπηρεσίας του Συμβουλίου. Δεν ξεκινάει αυτό κάποια κράτη-μέλη είναι μέσα στο κοινοτικό πλαίσιο, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ε, επικεφαλή. Οπότε δεν, δεν είναι κάθε φορά εξασφαλισμένη η παρακολούθηση, η εποπτεία. Σπάνια τα κράτη-μέλη δεν αποφασίζουν. Είναι και το θέμα της χρηματοδότησης. Δεν αποφασίζουν να είναι επικεφαλής κάποιο συγκεκριμένο κράτος. Οπότε όλα αυτά η συμμετοχή, όλα αυτά θα πρέπει κάπως να ρυθμιστούν και να αξιοποιηθούν καλύτερα. Άπαξ και Κοινοβούλιο και Κομισιόν ασχοληθούν και ε, ρυθμίσουν όλα αυτά. Πρόεδρε, συνάδελφε, σε αυτό το πνεύμα κινήθηκα κατά τη δουλειά μου μαζί βέβαια με τους σκιώδεις εισηγητές και ακριβώς όπως έκανε και ο Πασκάλ Λαντιρό ακριβώς όπως κάνουμε πάντα στην ε, Επιτροπή μας θα λάβουμε υπόψη ότι ιδέες, προτάσεις ε, εισφέρουν στη δουλειά μας οι συνάδελφοι. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Λαμασόγ. Να περάσουμε τώρα στους σκιώδες εισηγητές. Κυρία Μπρέσο δεν είναι εδώ, την εκπροσωπείτε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας μιλώ, όντως κύριε Λαμασούρ, εκ μέρους της Μερσέντες Μπρέσο. Λυπάται που δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά μου ζήτησε να σας διαβιβάσω τις εξής σκέψεις της. Η διαπίστωση της ε, πολυπλοκότητας για την υλοποίηση αυτής της ενσημένης εργασίας είναι σωστή. Θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη η χρησιμοποίηση αυτής της ενσημένης εργασίας, η πολιτική, να μην κατησχύει όσον αφορά το, ότι τα κράτη-μέλη θα χρειάζονται για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα να έχουν τέτοια συνεργασία και γενικώ η κυρία Μπρέσο συμφωνεί με τα προβλήματα που έχετε επισημάνει για την ενισχυμένη συνεργασία και συγκεκριμένα ε, η ομοφωνία που απαιτείται θεωρεί ότι είναι ένας φραγμός ότι δεν έχουμε κάποιο είδους ε, πάγιους κανόνες για τη διαχείριση, για την έναρξη, για τη, για τη λήξη της για τον ε, κίνδυνο, τα κράτη-μέλη να κινηθούν εκτός κοινοτικού δικαίου και να ε, εργαστούν, να κινηθούν σε διακυβερνητικό επίπεδο. Ε, η κυρία Μπρέσο επίσης θεωρεί ότι σε, αυτό, σε αυτή την έκθεση όπως και στην έκθεση Ντυρών έχουμε μια διαφοροποιημένη ολοκλήρωση και εκεί κάποιες υποκρατικές ε, οντότητες ότι θα πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν Βέβαια αυτό έχει και σχέση με το κατά πόσον το εθνικό δίκαιο τους ε, έχει απονείμει κάποιες νομοθετικές αρμοδιότητες Επίσης, ε, ε, όπως και εσείς κύριε Λαμασούρ, λέει κύριε Μπρέσο, ότι θα πρέπει να δούμε τον ρόλο, τον σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Κοινοβούλιο για αυτή τη διαδικασία. Επικαλούμεθα το άρθρο 225 γι' αυτό. Θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογη, άριστη η εκθεσή σας και έχει κάποιες προτάσεις που θα τις προτείνει ως τροπολογίες, ε, τις κατεβάσει ως τροπολογίες, ιδίως όσον αφορά την νομική βάση. Ε, θεωρεί το, ότι συντρέχει το τρόπο 25 και 352, ούτως ώστε να έχουμε τέτοιου είδους ε, λειτουργία και διαδικασία και επίσης για την αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων πρόκειται για ένα υβριδικό μέσο και γι' αυτό θα πρέπει να προσφύγει κανείς όχι μόνο στο κοινοτικό αλλά και στο εθνικό δίκαιο. Επίσης, λέει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συνεργασία και των τοπικών αρχών για διασυνοριακή ενισχυμένη συνεργασία. Ε, έχει εδώ σχέση και το τι κάνει η ΟΚΕ, η Επιτροπή των Περιφερειών. Αυτά από πλευρά της ε, κυρία ε, Μπρέσο. Βέβαια, σωστό είναι ότι λήφθη υπόψη το τι γίνεται, τι εμπειρίες υπάρχουν και έτσι τώρα θα πρέπει να καταλήξουμε στο να μην έχουμε δύο κατηγορίες κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Ούτε πρέπει να πούμε με συγκεκριμένο τρόπο τι θέματα μπορεί να περάσουν από αυτή την ε, συνεργασία, αλλά μέρα με τη μέρα προκύπτει αυτή η ανάγκη του ότι θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση των ε, ε, τοπικών, των περιφερειακών αρμοδιοτήτων και με κάποιο τρόπο να καταλήξουμε σε καλύτερη διοίκηση υπέρ επιχειρήσεων, υπέρ των πολιτών. Αυτό προκύπτει όλα ένα και πιο συχνά. Όλα ένα και πιο συχνά έχει, έχει ο κόσμος και η οικονομία παράπονα ε, για το ότι πολλές φορές η νομοθεσία αποτελεί φραγμό. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το καλύτερο αυτή η συνεργασία με δικούς της κανόνες και νομίζω ότι όλο ένα και περισσότερο θα χρησιμοποιείται. Άρα να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή έκθεση και έτσι να φτιάξουμε έναν ε, χάρτη πορείας όσο γίνεται καλύτερο. Ευχαριστούμε. Ως ε, σκιώδης ε, μέρος του ECR, να σας πω τα Αρχικά, μια σκέψη για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μόνο τους ε, ε, βουλευτές ε, που, από τις μετέχουσες χώρες που θα μπορούν να ψηφίσουν. Αυτό αντιβαίνει στην αρχή που έχουμε αυτή τη στιγμή για χώρες που δεν έχουν ευρώ, παρεμβαίνουν και ψηφίζουν στην Ολομέλεια για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ευρώ. Φαντάζομαι ότι θα το έχετε λάβει υπόψη αυτό. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε το σκεπτικό αυτής της διαφοράς μεταξύ των δύο πλαισίων, τη ενισχυμένη συνεργασία δηλαδή και των ε, τομέων ε, τη συνθήκη που δεν ισχύουν για κάποιε χώρε. Και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ένα επίτροπο θα πρέπει να έχει την πολιτική ευθύνη τη ενισχυμένη συνεργασία. Όμω έτσι δεν υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων, έστω ότι 10 χώρες ε, προχωρούν και 17-18 όχι μπορεί ο Επίτροπο να προέρχεται μία από, μία από τι χώρε που δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία. Και είναι το ηγετικό πρόσωπο. Εγώ θεωρώ και έχω την εντύπωση ότι ο Επίτροπο εκπροσωπεί όλα τα κρατημέλη, όχι μόνο ένα μέρο του. Αν θέσουμε λοιπόν ε, και δώσουμε αυτή την ιδιότητα στον Επίτροπο, μπορεί να δημιουργήσει και να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων. Τώρα, Κάποιος από την άλλη δεν θέλει να πάρει το λόγο. Χέλμουντ. Όχι. Πασκάλ. Παρακαλώ. Μάλιστα, πολύ σύντομα. Ο εκπρόσωπο δεν. Συγγνώμη, ο επίτροπο δεν εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη, αλλά το ευρύτερο ευρωπαϊκό συμφέρον. Επομένω, νομίζω ότι δεν υπάρχει ζήτημα σύγκρουση συμφερόντων για αυτό το φάκελο σίγουρα του κυρίου Λαμασού. Συμμερίζουμε σχεδόν στο ακέραιο την ε, θέση σας, όμως... Στο σημείο 18 θα ήθελα να πω κάτι για το διακοινοβουλευτικό σκέτο, σκέλος. Τα εθνικά κοινοβούλια που συμμετέχουν και το καθεξής. Εφόσον το εξετάζουμε στο πλαίσιο τη συνθήκη, έχουν να κάνουν με προπολογισμού που είναι εθνικοί, αλλά και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με, την ε, με τι αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαι επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Εδώ θα ήθελα να τα ξανασυζητήσουμε, αλλά σίγουρα όχι τώρα, γιατί τώρα θα ψηφίσουμε. Ε, thank you very... Ευχαριστούμε πολύ. Χέρερτ, ήθελες το λόγο. Όχι. Καστάλντο, όχι. So I, understand we can finish this point, and I would like to... Κλείνουμε λοιπόν αυτό το σημείο. can δεν θέλει κάποιο άλλο να πάρει το λόγο. Α, φυσικά, ο Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, για να μην καθυστερώ και τις ψηφοφορίες, να απαντήσω στους κοιόδες, λοιπόν και αυτούς που τους εκπροσωπούν. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και συμμερίζονται το γενικό πνεύμα ε, και τη συλλογιστική του σχεδίου έκθεσής μου. Για το χαραγή πρέπει να σας πω ότι για τις περιφέρειες πρέπει να λάβουμε υπόψη τις αρμοδιότητες που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη-μέλη νομοθετικής ε, φύσεως και έχουν εκχωρηθεί σε αυτές τις περιφέρειες. Πρέπει λοιπόν να δούμε. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι το κράτος μέλος και τα κάτι μέλη στο Συμβούλιο Υπουργών ε, εκφράσουν τον ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή σε αυτή την ενισχυμένη συνεργασία. Αυτή η συνεργασία μπορεί να σημάνει και την συμμετοχή και εμπλοκή ορισμένων περιφερειών και όχι κάποιων άλλων βέβαια. Ο κύριος Μέσερ Σμιτ μετά έθεσε δύο ερωτήματα. για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εάν υπάρχει ειδική επιτροπή ή διαρκής επιτροπή, αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε δικαίωμα ψήφου σε όλους όσοι συμμετείχαν μέχρι τώρα και πράγματι ισχύει αυτό κάθε φορά που ζητήσαμε για κάτι που αφορά την Ευρωζώνη. Μόνο λοιπόν σε αυτούς που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία πρέπει να τεθεί αυτό το ζήτημα και όπως προκύπτει από μία σειρά υποθέσεων και κρίσεων μεταξύ κρατών μέλων κάποια, τα τελευταία χρόνια, τι σημαίνει αυτή η θεμητή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και ένωσης. Στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας, όλα τα κατημέλη, όλοι οι ευρωβουλευτές, όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να ενημερώνονται και να συμμετέχουν, να έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν γνώμη, αλλά να μην έχουν την άμεση ή έμεση δυνατότητα ορισμένοι εκπρόσωποι ε, κρατών μελών να παρακολύσουν ε, την ενισχυμένη συνεργασία. Αυτό είναι ένα στοιχείο προβληματισμού, αλλά μπορούμε να βρούμε μια λύση για αυτό το ζήτημα. Για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Επιτρόπου που θα αναλάβει το φάκελο, ψήφισε, συγγνώμη, απάντησε και ο κύριος Διουγόν, αν είναι θέμα παιδείας, φυσικά και είναι επίτροπος παιδείας, γεωργίας και ούτω καθεξής, ανεξαρτήτως ε, της ε, εθνικότητάς του. Τέλος, ο Πασκάλ Ντιγόν μίλησε για την εθνική εκπροσώπηση στο πλαίσιο της, ε, του δημοκρατικού ελέγχου της ενισχυμένης συνεργασίας. Εξαρτάται από το θέμα. Εξορισμού πρόκειται μόνο για ζητήματα μεικτή αρμοδιότητα. Αν πρόκειται για αποκλειστική ε, αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε πολλέ περιπτώσει ε, είναι το Κοινοβούλιο, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμω, μετά από συζήτηση με τον πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπω ότι το δικαστήριο, όλο και περισσότερο, θα ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε τομείς που το δικαστήριο θεωρεί ότι είναι μεικτής αρμοδιότητας και που σε μεγάλο βαθμό στην πράξη είναι εθνικής αρμοδιότητας. Ό,τι έχει να κάνει με το οικογενειακό δίκαιο ή και το αστικό δίκαιο ευρύτερα. Αν έχουμε ψηφίσει και υιοθετήσει ενισχυμένη συνεργασία ε, για το δίκαιο που διέπει τα διαζύγια, τότε βλέπουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όμως αν πρόκειται για ε, ζητήματα Ευρωπαίων πολιτών που παντρεύονται σε άλλη χώρα και ούτε καθεξής, μετά υπάρχει ένα νομικό σκέλος και πολιτικό που δικαιολογεί την παρέμβαση της Ένωσης μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας και με τη σύμφωνη γνώμη του δικαστηρίου. Φαντάζομαι ότι μπορεί αυτό να ανατεχθεί και σε επίπεδο ποινικού δικαίου, όπου η κύρια αρμοδιότητα είναι σε εθνικό επίπεδο, τότε σε αυτήν την περίπτωση θεωρώ ε, λάθος ε, να αποτρέψουμε και να απαγορεύσουμε την εκπροσώπηση ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά και θα συναντηθώ και με τους ασκιώδες για να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά να σας ενημερώσω ότι προτείνεται να κατευθούν οι τροπολογίες μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Αν συμφωνείτε, αυτό θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε τις τροπολογίες στις 22 Ιανουαρίου και να περάσουμε στην ψηφοφορία στις 29 Ιανουαρίου και θα πάμε μετά στην Ολομέλεια. Το στομότερο δυνατόν. γιατί στο τέλος θα έχουμε καταβάσει τις νομοθετικές προτάσεις. Πρέπει λοιπόν ε, να το προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο νωρίς. Ωραία, κλείνουμε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Ας περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Αρχικά να ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε λοιπόν πρώτα ότι λειτουργούν όλα σωστά. Άρχεται η ψηφοφορία. One EPP too much. Ένας παραπάνω. One EPP is leaving, so all other EPPs have to vote. Φεύγει ένας, οπότε όλοι οι υπόλοιποι... Φεύγει ένας του ΕΛΚ. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να ψηφίσουν. Σας ευχαριστούμε. Η πρώτη ψηφοφορία θα γίνει για την πορεία τη συζήτηση για το μέλλον τη Ευρώπη. Ο εισηγητή Ραμόν Χαουρεγία Τόντο έχει δει στο λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δώστε μου λίγα λεπτάκια για να εξηγήσω στους συναδέλφους της Επιτροπής κάποια πράγματα σημαντικά. Πρώτα-πρώτα, να σας πω τι είδους έκθεση θα ψηφίσουμε τώρα. Υπενθυμίζω ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι εδώ να διατυπώσουμε γράφως αυτά τα οποία αποφασίσαμε τα τελευταία χρόνια και θέλουμε να υπάρχει κάποιο είδους ε, επικαιροποίηση μέσω των εκθέσεων ε, Verhofstadt, ε, Ressobrock και τι γίνεται κάθε φορά που έχουμε ακούσει από τους υπουργού στο Στρασβούργο οπότε τώρα έχουμε κάτι σαν χάρτη πορείας όσον αφορά το την πολιτική ζήμωση στο μέλλον και εξηγώ του τι δυνατότητες ξανοίγονται. Περί αυτού πρόκειται. Και βέβαια δεν καταλήγω σε συγκεκριμένες ε, λύσεις και προτάσεις. Απλώς σε γενικές γραμμές κατευθυντήριες φτιάχνουν έναν χάρτη πορείας τις βασικές κατευθύνσεις προς αντολισμούς για το μέλλον. Πρόκειται περί συνειδητικών προτάσεων και θα δείτε και από τις τροπολογίες που θα ψηφίσουμε ότι αυτό στο οποίο καταλήξαμε είναι οι αδρές γραμμές ε, κατανόησης συμφωνίας μεταξύ των πολιτικών πτερήγων του Κοινοβουλίου ε, εκείνων που θέλουν περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν θα έλεγα περισσότερη Ευρώπη θα έλεγα για μια Ευρώπη με καλύτερη ολοκλήρωση και το πνεύμα ε, είναι όλα αυτά που ακούσαμε και από πολλούς πρωθυπουργούς δηλαδή το ότι τα καταφέρνουμε καλύτερα όταν ενεργούμε από κοινού αυτά είναι η κεντρική ιδέα της έκθεσης δεν έχω κάποιες ε, κομματικές θέσεις περάσει εδώ γιατί συνοηθήκαμε με από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες και ολοκληρώνω ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον Έλμαν Μπρόκ του ΕΛΚ, την ε, Μάιτε Παγκάθ από τους φιλελεύθερους, τον Πασκάλ από τους Πρασίνους και την Μπάρβαρα Σπινέλη της ΓΚΟΕ. Τους ευχαριστώ για τη συνεργασία τους για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε αυτές τις αδρές γραμμές για μια καλύτερη Ευρώπη με καλύτερη ολοκλήρωση. Και όλες αυτές τις πολιτικές ομάδες αυτό το μήνυμα θα εκπέμψουμε τώρα μέσω της προεκλογικής ε, περίοδου για το τι πιστεύει το Κοινοβούλιο ότι πρέπει να γίνει. Έχουμε κάποιες ε, αρνητικές γνώμες σε διάφορες ε, συναρμόδιες επιτροπές όπως στην Ίντα, Άγκρι, Γιούρι, στην Κοντ. Αυτό γιατί προσπαθήσαμε σε κάποιες γενικόλογες παραγράφους να καλύψουμε τη δική τους θέση. Το, πνεύμα της ε, ε, γνώμη τους σε παραγράφους. Δεν κάτσαμε να κάνουμε ψηφορία για την κάθε παράγραφο χωριστά. Πάντως, η ΕΚΟΝ σε σχέση με αυτή την έκθεση ε, ενήργησε δυνάμει του άρθρου 54 του κανονισμού δηλαδή γνωμοδότησε ε, εμείς ε, αυτή τη γνωμοδότηση την ε, εντάξαμε στην έκθεση για να ξέρετε τι ψηφίζουμε και πάλι τις ευχαριστίες μου και συγγνώμη που έφαγα το χρόνο σας με αυτές τις επεξηγήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στη φοβορία η οποία θα διαρκέσει κάποιο χρόνο οπότε να παρακολουθείτε όλοι το τι σημαίνει. 68 λοιπόν, τροπολογία 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική β υπέρ, το L υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Α, όχι, τροπολογία 84. Δεύτερο τμήμα μόνο της 84 υπέρ. Κατά. Σοσιαστές είναι υπέρ. Καλώς. Εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική D υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές. Εγκρίνεται η συμβαστική η υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. F συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά το είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική H υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 113 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική I υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική, ε, όχι στη τζούρι 1, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική L υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, γιούρι 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 123 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική M υπέρ κατά αποχές έγκρινεται, συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική δέσμη έκον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 επόμενη τοπολογία σελίδα 17 υπέρ κατά να ελέγξουμε την τροπολογία 144 άρχεται η ψηφοφορία After all the colors of the compromises. It's 17. No, no, but, but if you go then, after the compromise, yes, exactly, so it's, it's 17. Σελίδα 17, λοιπόν, ξαναλέω, είναι η τροπολογία 144. Ψηφίζουμε ακόμα, δεν έχει ψηφίσει ένας συνάδελφος. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 154. Περιμένω τους συναδέλφους. Ο κύριος Μπόκερ ζητάει εκ νέου ε, να ψηφίσουμε για την τροπολογία 144. sorry colleagues did you find after the colours of the compromise on page we, have been voting Ολοκληρώσαμε, περάσαμε όλες εκείνες τις σελίδες, τις πολύχρωμες ε, με την συμβαστική τροπολογία και είμαστε στη σελίδα 17 με την τροπολογία 144. Ναι, Πρόεδρε, λέει ο κύριο Σόφλιν, ναι, το πρόβλημα για μας είναι στην δική μας λίστα ψηφοφορίας. Ε, η 144 βρίσκεται στη σελίδα 118. Ναι, λέει πρόεδρο, αλλά είπα ότι ψηφίζουμε τι 144, οπότε τελείωσε. 154 λοιπόν υπέρ. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Μπροκ.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 κατά αποχές απορρίπτεται 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 και 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική Q υπέρ ΕΛΚ καλώς κατά αποχές εγκρίνεται 190 στην επόμενη σελίδα 190 Τη βλέπετε όλοι. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε στην 194. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε στην ολική ψηφοφορία. Άγκρι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά, άγκρι 229 και πάλι εδώ επί όλων αυτών ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Για την ίντα τώρα. Και πάλι δέσμη υπέρ κατά αποχές έκρινεται. Μετά ψηφίζουμε δύο σελίδες πιο μετά ψηφοφορία ε, για τις τροπολογίες ε, A ως I της ίντα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται, συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Γιούρι 3 με σε τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Γιούρι 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Γιούρι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 227 υπέρ κατά Σοσιαλιστές είναι κατά. Καλώς απορρίπτεται. Συμβαστή δι υπέρ. Κατά. Συνολική και πάλι ψηφοφορία κόντε τώρα. Υπέρ. Κατά. Κατά. Εγκρίνεται. από κοινού ψηφοφορία κοντ, δηλαδή τροπολογία 1-16 και ούτω καθεξή. υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτεται. Συμβαστική x υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική p υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ κατά κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε σε αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά ελέγχουμε την τροπολογία 3, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 12 ψήφους υπέρ και 12 κατά. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά. Και πάλι τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 5 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 6 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται 7 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Z υπέρ κατά ελέγχουμε τη συμβαστική τροπολογία Z άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας.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 αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά οι σοσιαλιστές είναι κατά οπότε απορρίπτεται συμβαστική AB υπέρ συμβαστική λοιπόν υπέρ AB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκριση υπέρ κατά σοσιαλιστέ είναι κατά και το ΕΛΚ οπότε απορρίπτεται συμβαστική ΑΕ e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική AF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AI υπέρ κατά ελέγχουμε τη συμβαστική τροπολογία AI. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρασε της ψηφοφορίας απορρίπτεται με 12 ψήφους ε, κατά και 11 υπέρ. Οπότε ε, αψηφίζουμε και για την 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Από κοινού ψηφοφορία Agri BDE υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ψηφίζουμε επί του συνόλου της έκθεσης νομαστική ψηφοφορία ηλεκτρονικά, η ψηφοφορία. Closed. Πέραση της ψηφοφορίας και εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ και 6 κατά. Uh, Έχουμε τώρα την γνωμοδότηση του Μέσερ Σμιτ για το πρωτόκολλο του Οργανισμού του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά. Ας ελέξουμε την 3, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά. Το έλκτη ψηφίζει. Υπέρ. Κατά. Είστε υπέρ. Ωραία. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. I think it's adopted, but we check the same. We close the vote. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Question. Six in favor. Έξι Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά το ΕΛΚ είναι υπέρ ας ελέγξουμε τη 12 yeah, but I'm not sure. The vote is closed and it's adopted with the same majority, 16 to 8. Amendment 8. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία μονομαστική κλίση άρχεται. Uh, sorry, so the vote 22 to 2, it's congrat... Εγκρίνεται σε χαρητήρια στον εισηγητή. Now it's, Just now the statute. uh, dear colleagues, can we... Συνάδελφοι, ας ε, προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της μέσας διάταξης, η τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Can just do it. Uh, Those colleagues who want to stay, uh, please stay. Those who want to leave, please do it in... Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, παρακαλώ, με ησυχία. Σημείο 9, λοιπόν. Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. There is, there has been a request uh, from... Υπήρξε αίτημα του Γενικού Γραμματέα της ΕΤΕΠ προς το Συμβούλιο για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΤΕΠ το οποίο έτοιμα προωθήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη διαδικασία της διαβούλευσης και το βασικό στοιχείο της πρότασης έχει να κάνει με το Brexit. Λαμβάνει υπόψη τις ε, επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν τροποποιήσεις που έχουν να κάνουν με τον αριθμό των διοικητών, ε, το δικαίωμα ψήφου, το κεφάλαιο της ε, τράπεζας που προσαρμόζεται προς τα κάτω μετά την απώλεια ε, του μεριδίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχει και πρόταση αύξησης του αριθμού των αναπληρωματικών διοικητών και Έχουμε και την ε, παράταση του, ε, της ειδικής πλειοψηφίας ε, σε τρεις τομείς. Τα επιχειρησιακά σχέδια, τον διορισμό μελών της δικού σας επιτροπής και η υιοθέτηση του ιστορικού κανονισμού. Η πρόταση για την ΕΤΕΠ θεωρώ ότι χρήζει στήριξη, γι' αυτό το λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι τροποποιήσει αυτέ είναι σημαντικέ για τα κράτη-μέλη και για την εύρυθμη λειτουργία τη ΕΤΕΠ, ιδίω στο πλαίσιο του επερχόμενου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου και των δημοσιονομικών αναγκών. Σκοπός εδώ είναι και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της τράπεζας. Υπάρχει και μια πίεση χρόνου γιατί οι προτάσεις τροποποίησης θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ εγκαίρως, πριν δηλαδή από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το σημαντικό για την ΕΤΕΠ είναι να δείξει και στις αγορές ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη λειτουργία της. Είναι σημαντικό και για την ε, πολύ θετική αξιολόγηση της οποίας χαίρει η ΕΤΕΠ αυτή τη στιγμή και αυτό μεταφράζεται και στην τιμή του κεφαλαίου που εξασφαλίζει η ΕΤΕΠ από τις διεθνείς αγορές. Αρχικά, δεν ακολουθήθηκε η σωστή ε, διαδικασία. Είχε πάει σε λάθος επιτροπή. Τελικά αποφασίστηκε να την αναλάβει η ΑΦΚΟ. Δύο επιτροπές θα μπορούσαν να είχαν γνωμοδοτήσει, η Econ, η οποία όμως ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει ε, να γνωμοδοτήσει, και η Budget, η οποία ε, καταρχήν θέλει να δώσει γνωμοδότηση. Επιπλέον έχουμε και το θέμα της χρονικής συγκυρίας, του χρονοδιαγράμματος. Γι' αυτό θέλαμε να ακολουθηθεί η διαδικασία. Γι' αυτό και με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία θα ήθελα να προτείνω να εφαρμόσουμε μια απλουστευμένη διαδικασία με βάση τον κανόνα 50 του ιστορικού κανονισμού που ισχύει σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν τροπολογίες να περάσουμε σε ε, ταχεία υιοθέτηση. Μπορούμε λοιπόν να στείλουμε ε, την ε, έκθεση στην Ολομέλεια χωρίς τροπολογίες. Προτείνω λοιπόν ε, την απλουστευμένη διαδικασία δυνάμει του άρθρου 50. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους Σκιώδης. Αν θέλουν να πω κάτι, καμία πολιτική ομάδα δεν έχει μεταφέρει ονόματα σκιωδών προς τη γραμματεία. Εάν ισχύει λοιπόν αυτό, προτείνω το εξή. Όπω και να έχει, θα υπάρξει προθεσμία ε, κατάθεση τροπολογιών η 29η Νοεμβρίου στι 12 το μεσημέρι. να ψηφιστεί στις 6 Δεκεμβρίου στην ΑΦΚΟ για να περάσει την Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Εν τω μεταξύ ακόμα πρέπει να διευκρινίσουμε την κατάσταση με την ε, Επιτροπή Προπολογισμών, αν ε, δηλαδή την ικανοποιεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, προκειμένου και εμείς να κινηθούμε γρήγορα. βάσει της διαδικασίας της διαβούλευσης. Όπως προείπα, θα ψηφιστεί από την Επιτροπή μας στις 6 Δεκεμβρίου και θα πάει στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Εάν αλλάξει κάτι, θα σας ενημερώσω. Ωραία, κλείνουμε και αυτό το σημείο. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην ώρα μας σχεδόν στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης την ανταλλαγή απόψεων με μέλη της Επιτροπής από τις πλέον σημαντικές επιτροπές της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της Επιτροπής ΣΥΒΕΞ, Ιθαγένειας, Διακυβέρνησης, Θεσμικών και Εξωτερικών Υποθέσεων. σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.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 την πρόεδρο της Επιτροπής. And then we will proceed to the discussion. We will have, hopefully you, you are ready to do it, we should have one speaker per political group, which means that... Θα έχουμε έναν ομιλητή αναπολιτική ομάδα, επομένω πέντε συνολικά, από την Επιτροπή των Περιφερειών και 8 από την ΑΦΚΟ. Changes. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής. We'll have the, it organized the discussion um, this way, so I would like to, uh, to start, uh, we will correct the names and the list uh, in the... Λοιπόν, θα διορθώσουμε τον κατάλογο μελετών ε, στην πορεία. Πρώτα απ' όλα να δώσουμε το λόγο όμως στην κυρία Μπάρμπαρα Τούντεν. Δεν είναι εδώ ο κύριος Λάμπερ. I was thinking that, that as usual a woman is replacing the man, but it's not to do the job. I'm sorry, I just, nobody told me, I was, uh, okay, no, but... So... Συγγνώμη, δεν το είχα καταλάβει. Θέλετε να πάρει πρώτα το λόγο η κυρία Ντούντα. Ναι, ωραία. Και μετά ο πρόεδρος Χάιν Λάμπερτς. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Είδατε ότι εργαζόμαστε από κοινού με τον Καλ Χάινς και συνεχίζονται γερμανικά. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε Χούμπνερ και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και αγαπητοί συνάδελφοι της ΣΥΒΕΞ. Μετά από τις διμερείς συνομιλίες που είχαμε, κυρία Χούμπνερ, και μετά τον ενδιαφέροντα διάλογο που κάναμε με τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια τον Οκτώβριο, χαίρομαι πολύ που σήμερα βρίσκομαι εδώ για να συζητήσουμε λίγο πιο εντατικά αυτό το τόσο κεντρικό ζήτημα του μέλλοντος της Ευρώπης. Και ελπίζω πως θα δοθεί συνέχεια και θα ε, μπορούσε ενδεχομένω να θεσμοθετηθεί αυτό ο διάλογο και στα πλαίσια τη ανάληψη ε, των καθηκόντων του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή μετά από τι ε, ευρωεκλογέ. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χρήσιμο, δηλαδή να υπάρχει μια τέτοια τακτική συνάντηση με τα μέλη τη ε, ΣΥΒΕΞΕ. και έχετε ήδη δει πώ εμεί, ω εκπρόσωποι των αρχών τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να συμβάλλουμε στον διάλογο για το μέλλον τη Ευρώπη. Ε, μιλάμε για θεματικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία, τη σταθερότητα, τη βιωσιμότητα ε, και φυσικά υπάρχουν υπάρχει σωρία προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Τα όσα βιώνει η Ευρώπη κατά τις τελευταίες ε, δεκαετίες και χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο θεωρείται ως αυτονόητο αλλά ε, απειλείται έξω ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, τα δικαιώματα των ε, μειονοτήτων αλλά τελικά και τα δικά μας τα προστοζέν. Εμείς λοιπόν ε, ως θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφορετικές αρμοδιότητες αλλά στενά συνδεδεμένα, ε, μεταξύ τους, ε, συνδεδεμένες μεταξύ τους ε, θα πρέπει ειδικότερα και στο πλαίσιο της καλύτερης διακυβέρνησης να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Επιτροπή των Συνταγματικών Υποθέσεων της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει πρεσβεύσει επανειλημμένα πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες εδώ ε, και ε, η πρόσφατη έκθεση του συναδέλφου Αντωνίου Εντήλ πραγματικά συμπεριλαμβάνει μια σειρά από πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία υποστηρίζουμε και εμείς ειδικότερα σε ό,τι αφορά το να καταστεί πιο διαφανής ο τρόπος εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ένωσης γιατί με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να διασφαλίσουμε υψηλότερη αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων και προκειμένου βέβαια με αυτόν τον τρόπο να καταστήσουμε την ε, δημοκρατία πιο ζωντανή ε, και πιο εύρωστη ε, για να αντιμετωπίσουμε και τους εχθρούς της. Ωστόσο, τα όσα διαπιστώνουμε δείχνουν ότι ακόμα θα πρέπει να πείσουμε για πολλά περισσότερα ακόμα του πολίτε μα. Εμεί από την πλευρά ε, τη Επιτροπή Σύμβεξη, τη Επιτροπή των Περιφερειών, δεν ασχολούμαστε μόνο με ζητήματα διακυβέρνηση, αλλά και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ε, μετανάστευση, εξωτερικών σχέσεων και άλλα. Άρα λοιπόν εμεί ε, θεωρούμε στην πλειοψηφία μα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει περισσότερε αρμοδιότητε έτσι ώστε οι πολίτε να αναγνωρίσουν και να βιώσουν περισσότερο την αμοιβαία του συνεργασία και την αλληλεγγύη του. Ε, αυτό τι σημαίνει σε επίπεδο δημοκρατίας ε, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα να υπάρχει βούληση προς αυτή την κατεύθυνση, ε, να υπάρχει άλληλο σεβασμός και βούληση για την εξέβρεση κοινών λύσεων. Και εδώ έρχομαι σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στον τομέα της διακυβέρνησης, το οποίο θα ήθελα να σας θέσω σε ό,τι αφορά και αυτή την έκθεση και μελλοντικέ εκθέσεις, αλλά και το μέλλον γενικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βασίζεται στην πολυμορφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στις ε, διάφορες περιοχές της, περιφέρειές της, τις πόλεις της και τους ε, πολιτισμούς και τις κουλτούρες τους, τις οποίες θα πρέπει να διατηρήσουμε. Και γι' αυτό λοιπόν κατά τη δική μας άποψη ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών αυτοδιοίκηση είναι σημαντικό στο πλαίσιο δηλαδή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπως θα ακουστεί και μέσα στη συζήτηση τώρα. Δηλαδή, η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνηση δεν είναι τόσο τεχνική όσο ακούγεται. Ε, σημαίνει ότι όλα τα επίπεδα τη διακυβέρνηση θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ του, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα, την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή, αλλά και τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, αυτή η έννοια θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλα τα κείμενα για το μέλλον τη Ευρώπη, αλλά να λαμβάνεται και υπόψη σε όλε τι μελλοντικέ προτάσει για τη μεταρρύθμιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτου ε, δικαίου θα πρέπει πάντοτε να τη χάνουν σεβασμού και ε, μια αντίστοιχη ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, για τη διαχείριση τη μετανάστευση και η έλλειψή τη αυτή τη στιγμή ε, γίνεται αισθητή ακριβώ στι δικέ μα περιφέρειε γιατί ακριβώ οδηγεί σε μία μείωση τη αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων τη Ένωση, πράγμα το οποίο με τη σειρά του στο πλαίσιο των εκλογών οδηγεί στην ανάδυση λαϊκιστικών δυνάμεων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, διαδικασίες οι οποίες θα επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα, στα, στα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει εμπλοκή ακριβώς των τοπικών και περιφερειακών ε, αρχών προκειμένου να τραφεί περισσότερο από αυτές τις διαδικασίες η, η δημοκρατική διαδικασία. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στη δημοκρατία και να ανοιγοδομήσουμε, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη τους στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Εμείς στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ε, θα είμαστε εταίροι σας και σας ευχαριστώ πολύ για την ε, δυνατότητα που μου δώσατε να παρέμβω σήμερα εδώ. Εμείς ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και για την εκδήλωση με τα Εθνικά Κοινοβούλια που ήρθατε πριν από κάποιες εβδομάδες και μίλησαμε για τους Ευρωπαίους, για τη διαφάνεια, για το μέλλον της Ευρώπης. Και υπάρχει και σχετική γνωμοδότηση που έχει εγκριθεί στην Επιτροπή των Περιφερειών. Και πάλι, καλώς ορίσατε. Έχετε τον λόγο. κύριος Πρώτα πρώτα, κυρία Χιούμπνερ, κάτι που είναι μια ανάμνηση μας πολύ θετική και είναι η πάρα πολύ καλή ε, συνεργασία που είχαμε τότε που είχατε το χαρτοφυλάκι ως Επίτροπος της Περιφερειακής Πολιτικής. Με τέτοια ε, μικρά παραδείγματα που δείχνει την υποστήμενη αξία της η Ευρώπη. Πολύ πολύ όμορφη ανάμνησή μου είναι αυτή και προδικάζει και το μέλλον σίγουρα. Οπότε θα ήθελα να αρχίσω με κάποια απλή αλλά σημαντική διαπίστωση. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών είναι ερετή. Και αυτό ισχύει και σε τοπικό επίπεδο. Και ακριβώς όπως μέλη του Κοινοβουλίου είναι κάποιοι που έχουν εκλεγεί και κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό τη σήμερα ημέρα ότι και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ασχολούνται με τα προβλήματα επιτόπου και θεωρούνται εκπρόσωποι των Ευρωπαίων, οι βουλευτές και τα μέλη. Ε, εκείνοι τελικά κρίνουν το πώς θα δημορφωθεί αύριο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά ο κόσμος θα το κρίνει ε, και Αυτούς πρέπει να πείσει κανείς για όλα αυτά τα θέματα. Είναι ο ρόλος αυτός των ε, ερετών ε, μελών που έχουν να παίξουν αυτόν τον ρόλο στην επανίδρυση της Ευρώπης. Και γι' αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει οι δεσμοί μας να συσφιχθούν. Ε, είναι ταραγμένη η καιρή μας, η ευρωπαϊκή οικοδόμηση ποτέ δεν ήταν ένα ταξίδι στην Νινεμία, αλλά θα πρέπει τώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι τα όσα γίνονται είναι πάρα πολύ έντονα και επομένως θα πρέπει με λογική και με ε, ευθύτητα κανείς να κινηθεί μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια και όποιος λέει όχι στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία ε, επιτίθεται σε δικαιοσύνη, επιτίθεται σε μέσα ενημέρωση, λένε ότι η Ευρώπη είναι η ενσάρκωση του κακού. Ε, θα πρέπει αυτά με ευφυΐα να τα αντιμετωπίσουμε. Πολύ σημαντική η συζήτησή σας για το μέλλον της Ένωσης και αν κατάλαβα καλά ε, εγκρίνεται τη σχετική ε, γνωμοδότηση. Και είδα από το σχέδιο που διάβασα ότι στο κείμενό σας λέτε αυτά που και εμείς τονίζουμε στη δική μας γνωμοδότηση. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά η ουσία του μηνύματος είναι η ίδια και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και όσον αφορά τη ζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με τους πολίτες διάλογος με τους πολίτες. Πολλές φορές οι πολίτες δεν ξέρουν τι, να, τι να κάνουν, πώς να ενεργήσουν. Είναι σημαντική αυτή η φάση, είναι φάση προεκλογική. Όλα όσα γίνονται τώρα καλά είναι, αλλά ο αυθεντικός διάλογος δεν θα πρέπει να σταματάει στις εκλογές. Και από πλευρά μα έχουμε αυτή τη γνωμοδότηση του Οκτωβρίου και το μέλλον τη Ευρώπη Γίνανε πολλέ συζητήσει, ε, έρευνες, μελέτες, επιστημονικές. Αυτά από πάντοτε βοηθούν εμάς τους ε, πολιτικούς μας, ε, τεκμηρώνουν αυτά που λέμε. Όμως, πολλά λέγονται σε όλες τις χώρες Υπάρχει υποστήριξη προς την Ευρώπη, αλλά όχι αρκετή για να είμαστε ικανοποιημένοι. Εγώ δεν είμαι ε, ευχαριστημένο. μια που έχουμε ένα τρίτο των Ευρωπαίων που είναι κατά της Ένωσης. Και οι ανησυχίε του κόσμου αφορούν τα καθημερινά θέματα, απεργία, μετανάστευση, τα κοινωνικο-οικονομικά, και πάρα πολύ επίσης θεωρούν πάρα πολύ σημαντική την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μέσα σε ένα κόσμο όλο ένα πιο εγωιστικό οπότε και θεωρώ βέβαια ότι υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης. Έχουμε τρεις άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθούμε. Πρώτα πρώτα συχνά θεωρούμε ότι έχει δύο διαστάσεις η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Αυτό που εσείς ενσαρκώνετε, την διάσταση την ενωσιακή και από την άλλη μεριά η διάσταση που αφορά τα κράτη-μέλη. Όμως νομίζω ότι υπάρχει και μια τρίτη διάσταση, δηλαδή οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδων οργάνων φορέων και εκεί οι αιρετοί άρχοντες ε, βρίσκονται σε επαφή με τους Ευρωπαίους και αυτό είναι πλούτος τεράστιος 100.000 ε, κοινότητες, 300 περιφέρειες και χιλιάδες επίσης ενδιαμέσων φορέων. Αυτός ο πλούτος θα πρέπει να τύχει εκμετάλλευσης περισσότερες και να ξανάρθει κοντά σε αυτά όλα ο πολίτης. Θα πρέπει να εμπλακούν οι περιφέρειες και οι πόλεις στην ε, οικοδόμηση της Ευρώπης. Να μην είναι απλοί παρατηρητές εκτελεστικών κινήσεων. Υπάρχουν ε, πολλές, πάρα πολλές δυνατότητες. Αυτό το επιβεβαιώνουν οι πολίτες. Το, το λένε οι έρευνες που γίνονται, το ευρωβαρόμετρο. Το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο πιστεύονται περισσότερο από όλα τα άλλα επίπεδα διακυβέρνησης. Περισσότερο από το γνωσιακό το ευρωπαϊκό. Άλλη παρατήρηση θα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις εκεί που πρέπει, στο επίπεδο που πρέπει, και όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες. Αυτό θα πει επικουρικότητα. Πού το, το ξέρετε αυτό, όπω το ξέρουμε και εμείς. Πρόκειται για ε, μία έννοια που μας βοηθάει να προοδεύσουμε, να προχωρήσουμε. Ε, σε κάποιο είδους ε, αρνητικές, όχι επικοδομητικές εκδηλώσεις στο Κοινοβούλιο. Όχι, χρειάζεται κάτι πιο πλήρες, πιο επικοδομητικό, πιο αποτελεσματικό. Όλοι οι οποίοι ε, σχετίζονται με την νεολαία θα πρέπει να κινούνται έτσι επικοδομητικά όχι με μικροπολιτικές εκδηλώσεις. Και θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και η έννοια της επικουρικότητας, γιατί πολλές φορές η επικουρικότητα χρησιμοποιείται ως όπλο κατά της Ένωσης. Λένε ότι θα πρέπει να δώσουμε όσο είναι λιγότερες αρμόδιες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κρατήσουμε εμείς, μα δεν είναι αυτό. Θέμα δεν είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί στο δικό της επίπεδο και τα υπόλοιπα στο επίπεδο που αρμόζει, που αποδίδει. Άρα δεν είναι θέμα ε, μεταδίδας αρμοδιοτήτων, είναι πολλές φορές η, η πολυνομία. Αυτά θα πρέπει να δούμε με κριτικό μάτι. Τρίτη παρατήρηση, να συνεχίσουμε να φέρνουμε τον κόσμο κοντά στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βλέπουν το ότι υπάρχει αμφίδρομη σχέση. Όσο συμμετέχουν, ό,τι λένε οι Ευρωπαίοι, αυτό είναι κάτι το οποίο επιστρέφει σε αυτούς. Ό,τι κάνουν επίσης επιστρέψουν. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να το διακρίνει συνέπεια. Η ΟΚΕ, η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελούν ένα βήμα όπου όλα αυτά τα επεξεργαζόμαστε, όλα αυτά τα δημιουργούμε για να καταλήξουμε σε αποτελεσματικότητα σε κάθε θεσμικό όργανο. Και, εν κατακλείδη, να σας πω ένα πράγμα το οποίο πολλές φορές μας ε, διαιρεί. Πρόκειται φυσικά για τα οικονομικά. Ποτέ δεν τα καταφέρουμε χωρίς ε, πρικοδότηση και δεν αρκεί να δείχνουμε τον προπολογισμό και να λέμε όλα τέλεια. Χρειάζεται επαρκή προπολογισμό. Αλλιώ δεν μπορεί να οικοδομηθεί η Ευρώπη. Και είμαστε 300% υπέρ των όσων λέτε εσείς για το 1,3 του ΑΕΠ των κρατών μελών και ξέρουμε όπως και εσείς τι δυσκολίες υπάρχουν για την υλοποίηση αυτού του στόχου από πλευράς του Συμβουλίου εμείς σας υποστηρίζουμε, αλλά τη μάχη θα τη δώσετε εσείς. Δεν αρκούν οι 100.000 δήμοι και που εκπροσωπούμε για το Συμβούλιο και συγκεκριμένα για τους υπουργού Οικονομικών. Άρα και στο μέλλον αυτό ισχύει για τον προϋπολογισμό. Ε, επίσης, η πολιτική της συνοχής είναι κάτι που βγαίνει κατευθείαν από το DNA της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και θέλουμε την επόμενη εβδομάδα να ολοκληρώσουμε το έργο μας όσον αφορά όλες τις προτάσεις κανονισμών που συζητούμε και νομίζω ότι είναι τώρα η σωστή ώρα γιατί δεν ωφελεί κανείς να τα διαβάζει ούτε ωφελούν οι γνωμοδοτήσεις μετά την απόφαση. Γι' αυτό σας λένε, επόμενη εβδομάδα έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να κάνουμε και να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία για την λήψη αποφάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε για την παρέμβασή σας. Εδώ θα βρείτε πολλούς που θα υποστηρίξουν το μήνυμά σας, αλλά να σας πω ότι του χρόνου έχουμε χρονιά εκλογών. Σε πολλά κράτη-μέλη, εμείς ως υποψήφοι αυτών των εκλογών, συχνά είμαστε οι μόνοι που συμμετέχουν στην προεκλογική εκστρατεία, μιλούμε για την Ευρώπη και τελικά μας βλέπουν σαν ε, αυτούς που έρχονται κατά καιρού και μιλούν για την Ευρώπη στους πολίτες. Ελπίζω αυτή τη φορά και τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και τα μέλη της Επιτροπής σας ε, να δουλέψουν μαζί μας αυτή την προσπάθεια. Γιατί αυτή τη φορά πραγματικά πρόκειται για μία μάχη για το μέλλον της Ευρώπης. Είπατε και εσείς ότι η δημοκρατία δεν έχει να κάνει μόνο με τις εκλογές. Οι εκλογές είναι ένα κομμάτι της δημοκρατίας, αν και πολύ σημαντικό στοιχείο. Πριν από την αφήξή σας, σήμερα είχαμε δύο σημαντικές ε, εκδηλώσεις. Είχαμε εκπροσώπηση νέων Ευρωπαίων πολιτών που ήρθαν στο Κοινοβούλιο για να μας ε, που είχαν έρθει τον Ιούνιο στο Κοινοβούλιο για να μας μιλήσουν ξαναήρθαν ναι, τώρα, μας μίλησαν για την Ευρώπη και τις ιδέες τους. Ένας από την Ουγγαρία, ένας, μία από την ε, φύρα που ελπίζουμε σύντομα να αποκαλείται Μακεδονία και ένας τρίτος Γερμανοβούλγαρος και Ευρωπαίος όπως δήλωνα. Μας βοήθησαν να κατανοήσουμε και τις προτάσεις και τις ιδέες και τις προσδοκίες τους. Και είχαμε και την έκθεση Χαουρέγγι. η οποία εγκρίθηκε και αυτό είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Να δώσω το λόγο στο Ραμόν, λοιπόν για να μας μιλήσει όχι μόνο για την έκθεση, αλλά και για την ουσία της. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χαρούγι. Να σας τα πω στα ισπανικά. The audio. Βάλτε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μου δίνετε το λόγο ούτως ώστε μαζί με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας να σας πω σχετικά με την ψηφορία μας ότι αποφασίσαμε όπως γνωρίζετε και όπως ήδη σχολιάσατε ε, έχουμε αυτήν την ε, έκθεση για το μέλλον της Ευρώπης και έτσι θέλαμε να ρίξουμε φως στις διαφορετικές προτάσεις όλων των πολιτικών ομάδων αλλά την ΚΟΖΑΚ, την ε, ε Επιτροπή των Περιφερειών, την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Πρόκειται για ένα συνεχή διάλογο, μια συνεχή προβληματική για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Είναι τώρα περίπλοκα τα πράγματα για την Ένωση. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι κάπως μπερδεμένη, περίπλοκη αυτή η περίοδος. Και η γνωμοδότηση που εγκρίναμε χαράζει κάποιες ε, βασικές κατευθυντήρες για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Και τονίζω το πόσο σημαντικό είναι το ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών ε, θέλουν να κάνει βήματα πρόοδου η Ένωση. Είναι κάποιες ενέργειες κατεπίγονωσες που πρέπει να γίνουν για το μέλλον της Ένωσης για την άμυνα, για την εξωτερική πολιτική, για την διακυβέρνηση της ε, ΟΝΕ, για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, για την ε, μεταναστευτική πολιτική, για όλες αυτές τις σπουδαίες ε, προκλήσεις. Η έκθεση αποτελεί χάρτη πορείας. με τώρα ναι. το ότι θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική η Ευρώπη να έχει περισσότερη ολοκλήρωση για να πετύχει την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Και είναι τώρα το θέμα επίσης της κατανομής ανομοδιοτήτων μεταξύ των ομοκέντρων κύκλων ε, αυτών που ε, έχει ένωση τοπικό επίπεδο, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και Υπάρχει συμφωνία στο ότι αυτές οι μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα και της παγκοσμιοποίηση απαιτούν η Ευρώπη να έχει την δυνατότητα να κάνει καλύτερα τα πράγματα αυτά που τα κάνουμε μαζί από κοινού. Αυτή είναι η ιδέα που κυριαρχεί ε, στην κουβέντα, στην προβληματική που ισχύει εδώ στο Κοινοβούλιο. Και έχουμε επίσης τις επικουρικές ε, λειτουργίες αυτές του που αφορούν την, ε, το περιφερειακό επίπεδο και το τοπικό επίπεδο, ότι δηλαδή αυτά μπορούν να γίνουν εκεί, θα πρέπει να γίνονται εκεί. Και αυτό ε, γίνεται σεβαστό. Επίσης, θα πρέπει να συζητηθούν κάποια προβλήματα και αυτά να τα συζητήσουμε μαζί, μαζί με εσά. Πώς θα έχουμε καλύτερη συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά την καθημερινή διοίκηση, διακυβέρνηση. Πώς πιο αποτελεσματικά θα μεταφέρουμε την φωνή των περιφερειακών, των τοπικών αρχών που δίνουν τεράστιες δυνατότητες για επαφή του κόσμου με τα θεσμικά όργανα. Πώς αυτό, αυτή η λειτουργία θα είναι καλύτερη. Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο. Αυτά που εκφράζουν οι περιφέρειες στο πλαίσιο της διακυβέρνησης και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι στην Επιτροπή Περιφερειών αναφέρονται τα προβλήματα για τις περιφέρειες που έχουν ευρείες νομοθετικές ε, αρμοδιότητες και ε, ακούγεται και η φωνή των περιφερειών που δεν έχουν τέτοιες αρμοδιότητες. Ε, οπότε υπάρχουν αυτές οι σημαντικές διαφορές όπως γνωρίζουμε στις εθνικές ε, δομές λειτουργίας υπάρχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα ε, αρμοδιοτήτων νομοθετικών. Οπότε οι περιφέρειες που έχουν τέτοιες αρμοδιότητες ζητούν μεγαλύτερη παρουσία των υπολείπων που δεν έχουν ακόμα νομοθετικές αρμοδιότητες. Επομένως, θα πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός των εθνικών ε, δραστηριοτήτων και ισόφιλος των πολιτών αυτές οι αρμοδιότητες παρουσιάζουν προβλήματα και φραγμούς σε επιχειρήσεις και σε Ευρωπαίους. Αυτά είναι τα τρία θέματα που θέλω να σας θέσω. Η Επιτροπή των Περιφερειών, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει όλο ένα και περισσότερο να είναι ισχυρότερη και να έχει ρόλο όλο ένα και πιο δεσμευτικό στην νομοθετική λειτουργία της Ένωσης. Ευχαριστούμε. Τώρα φτάσαμε στο τέλος ε, της γεναδορίας μου πλευράς ε, χρόνου. Πρέπει πλέον ε, να εφαρμόσουμε ένα χρονικό όριο των δύο λεπτών για να πάρουν όλοι το λόγο. Ο Έλμαρ Μπρόκ θα πάρει πρώτος το λόγο γιατί πρέπει να αποχωρήσει. Και μετά ο κύριος ε, Αμπραμιβίτσιους. Έλμαρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, αγαπητέ Καλχάιντς, χαίρομαι που βρίσκεσαι ε, εδώ και γνωρίζεις πόσο μου αρέσει που κάνουμε μια τέτοια συζήτηση γιατί πραγματικά ο ο ρόλος εδώ που παίζει η Επιτροπή των Περιφερειών ως εκπρόσωπος των αρχών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι πραγματικά κεντρικός όπως έχει ήδη τονιστεί από δική μας πλευρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό επιχαίρω ε, το σχόλιο που κάνατε ότι δηλαδή με τη δική σας δουλειά ουσιαστικά μπορείτε πραγματικά να τροφοδοτήσετε και να συμβάλλετε στη δουλειά που, που κάνουν οι συγγητές μας, ε, ούτω ώστε πραγματικά πάντοτε να λαμβάνετε περισσότερο η υπόψη της, ε, η άποψη της Επιτροπής των Περιφερειών γιατί αν δεν το κάνουμε, αν δεν τη λαμβάνουμε υπόψη θα χάσουμε πολλά. Ε, και αυτό βέβαια εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια που κάνουμε προκειμένου να ε, βρει και περισσότερη απήχηση η Ευρωπαϊκή Ένωση στις πατρίδες μας. Γιατί βέβαια αυτό είναι και το πρόβλημα, ότι αυτή η υπερβολική γραφει... γραφειοκρατικοποίηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντοτε γίνεται πάρα πολύ αισθητή και τονίζεται από, τις, από αυτές τις αρχές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και δεν θέλουμε να προβάλλουμε με τέτοιο τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα ακόμα γενικό σχόλιο. που αναφέρθηκε από την κυρία Αντούνα και από τον ε, κύριο Λάμπερτ σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη ταυτότητα και ούτω καθεξή. Αυτό βέβαια αποτελεί ένα ζήτημα του πώ μπορούμε να υπερασπίσουμε ε, την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση απέναντι στου εθνικιστέ. Οι εθνικιστέ, και εδώ δεν θα αναφερθώ στα ζητήματα παγκοσμιοποίηση και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αυτοί θεωρούν, πάντω φρονούν πω το βασικό ζητούμενο για αυτού, το σημείο αναφορά, είναι το κράτο. Ζητώ συγγνώμη, από το γραφείο μου πρέπει να είναι. Πάντοτε τα καταφέρω να παίρνω τηλέφωνο όταν έχω πάρει το λόγο. Συνεχίζω λοιπόν. Ε, θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να καταφέρουμε το εξής. Η κατανόηση η δική μου που έχω του κράτους είναι περιφέρειες από τη μία πλευρά και μετά ομοσπονδιακό κεντρικό κράτος. Ε, ένα τέτοιο σύστημα βέβαια και μια τέτοια παράδοση δεν ισχύει σε όλα ε, τα κράτη-μέλη. Αλλά με αυτόν τον τρόπο αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν θέλει κανείς ε, πραγματικά να είναι πεπισμένο σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα, ως Ευρωπαίος δηλαδή πολίτης, τότε θα πρέπει να υιοθετεί ταυτόχρονα με την εθνική του ταυτότητα και την ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή του ταυτότητα και είχε πει και κάποτε ένας ε, επιφανής ε, ε, Γερμανός ότι η δική μου γενέτειρα είναι η τάδε πόλη, η Γερμανία είναι η πατρίδα μου και το μέλλον μου είναι η Ευρώπη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνενώσουμε αυτές τις ταυτότητες έτσι ώστε η Ένωση πραγματικά να γίνεται αισθητή και στους πολίτες στο πλαίσιο και αυτής της πολυμορφίας που έχει της γλωσσικής, της πολιτισμικής και ούτω καθεξής η κεντρική Ευρώπη όταν ε, ε, ε, γίνεται αντιληπτή ως κεντρική θα αποτύχει γιατί οι πολίτες δεν απευθύνονται στην κεντρική Ευρώπη ακριβώς επειδή φοβούνται πως θα απολέσουν την ταυτότητά τους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προφάλουμε και πάλι ακριβώς αυτήν την, τις πολλαπλές ταυτότητες που μπορεί να έχει ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, λέει κύριο Πρόεδρο, ε, τον κύριο Αμπραμαβίτσιο, δίνω τώρα το λόγο. Ζητώ συγγνώμη που σα διακόπτω. Απλά ενημερώνω του συναδέλφου ότι υπάρχει web streaming, ε, δηλαδή μα παρακολουθούν ζωντανά. Ε, σα ενημερώνω απλώ όλου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ κάποια σχόλια από την πλευρά του ΕΛΚ και να πω ότι σε ό,τι αφορά σύμπαν τη Ευρώπη για του ε, πολίτε, θα πρέπει πράγματι να ε, ενισχύσουμε τι δυνατότητε συμμετοχή ε, των πολιτών και να έχουμε δυνατότητε μονίμου διαλόγου με του πολίτε. Και αυτό για την περίοδο μετά από το 2019. Αυτό είναι σημαντικό για να αυξηθεί η δημοκρατική νομιμότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και προκειμένου να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκύτερα στου πολίτε. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό όραμα, δίνοντα ε, την εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να λαμβάνει δράσεις πάντοτε σεβόμενη τις αρχές της επικουρικότητας. Ε, και βέβαια θα πρέπει να διευκολύνουμε όπως είπα και τις δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νόμιμο μια νόμιμη δομή διαλόγου με τους ε, πολίτες ε, στην οποία θα συμμετέχουν και τα θεσμικά όργανα. Ε, και η δική μας πολιτική ομάδα, το ΕΛΚ και από κοινού με την Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνουν ένα τέτοιο είδους διαλόγου και με τις τοπικές κοινότητες. Γιατί πολλές, πολλά είναι τα ερωτήματα και μάλιστα καινοτόμα που μας θέτουν ε, αυτές οι τοπικές κοινότητες. Για παράδειγμα στη Λιθουανία, πατρίδα μου δηλαδή, συζητείται πολύ το ζήτημα της ε, μελλοντική άμυνας και ασφάλειας. Ε, πρόκειται δηλαδή για ένα νέο στοιχείο πολιτικής. Επίσης υπάρχουν πολλοί ε, πολίτες οι οποίοι θέτουν ερωτήματα σε ό,τι αφορά την οικονομική στρατηγική της Ένωσης. Γιατί δεν είναι όλα ζητήματα που εντάσσονται στη λογική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Υπάρχουν και περαιτέρω θέματα. Άρα λοιπόν, νομίζω πως σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή των Περιφερειών που εκπροσωπεί ακριβώς αυτές τις ε, αρχές, τις τοπικές και περιφερειακές, ε, βρίσκεται στο πλευρό ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακριβώς στον στόχο αυτό της αύξησης δηλαδή της κοινωνικής συμμετοχής της αναγού συμμετοχής από την πλευρά των πολιτών προσπαθώντας ακριβώς να καταδείξει την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια σειρά από τομείς όπως η ασφάλεια και η άμυνα όπως η δημοκρατία όπως το κράτος δικαίου. Ε, νομίζω λοιπόν πως το σλόγγαν μας, το σύνθημά μας ε, για τις επόμενες ευρωεκλογέ θα πρέπει να είναι ε, «Η Ευρώπη είναι το μέλλον μας». Και το περιεχόμενο που θα δώσουμε σε αυτό το σύνθημα είναι κάτι το οποίο θα το καθορίσουμε εμείς οι ίδιοι. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για τους σοσιαλιστές τώρα, η κυρία Ιζόντερης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πώς θα καταφέρουμε να μας εμπιστεύονται και πάλι οι πολίτες μας. Δεν θα το καταφέρουμε αν ε, αναφερόμαστε μόνο στο Brexit και στον εθνικισμό. Αλλά αυτά συζητώνται ή τουλάχιστον αυτά εκλαμβάνουν οι πολίτε που συζητώνται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και βέβαια δεν θα πρέπει μόνο να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι γενικέ κοινωνικέ συνθήκε θα πρέπει να είναι και αυτέ οι κατάλληλε. Άρα λοιπόν το να επαναπροσανατολιστούμε και πάλι στην κοινωνική Ευρώπη είναι σωστή ε, άγουσα. Γιατί ήδη καταφέραμε κάποια ε, πράγματα, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και τις συνθήκες εργασίας και η νέα ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασία, η οποία θα δημιουργηθεί τώρα από τον Ιανουάριο του 2019, ε, αλλά ε, και αυτό το ζήτημα τη σύγκριση, δηλαδή τη ισότητα των μισθών στο ίδιο σημείο εργασία, αλλά και η υιοθέτηση τη νέα οδηγία σε ό,τι αφορά την απόσπαση των εργαζομένων, όλα αυτά αποτελούν τρόπου για να επιτύχουμε ακριβώ την πρόληψη του κοινωνικού ντάμπινγκ. Αλλά το να έχουμε μία σειρά από διατάξει δεν επαρκεί από μόνο του. Πρέπει να δώσουμε σάρκα και ωστά στην κοινωνική ε, πολιτική μας. Δηλαδή αν θέλουμε πραγματικά μια κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη θα πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο ε, ελάχιστο μισθό το οποίο για παράδειγμα θα βασίζεται στον, ε, στο μέσο όρο των μισθών ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ένα ελάχιστο μισθό, το κατώτερο εισόδημα θα πρέπει πραγματικά να ανταποκρίνεται σε ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωση, έτσι ώστε ο κάθε Ευρωπα... Ευρωπαίο πολίτη να νιώθει ασφαλή. Αποτελεί λοιπόν ένα τέτοιο ελάχιστο μισθό το καλύτερο όπλο μα στην καταπολέμηση τη ε, φτώχεια. Και εδώ βέβαια με απασχολεί ιδιαίτερα και η προστασία και τη δημοκρασία ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν μπορούμε να αμφισβητούμε και να θέτουμε ένα αμφιβόλο τη, δημοκρατικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώ επειδή οι ε, πολίτε μα. Ε, φοβούνται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να του ε, δώσουμε και πάλι αυτή την ασφάλεια που θα νιώθουν σε ό,τι αφορά τη διαβίωσή του. Ε, και επίση ε, επιτρέψτε να αναφερθώ και στο ζήτημα τη αλληλεγγύη, γιατί και αυτό τώρα βρίσκεται σε κίνδυνο. Δηλαδή πολλά κράτη-μέλη θέτουν προτεραιότητε εθνικέ πάντοτε και του δίνουν προτεραιότητα έναντι των ευρωπαϊκών. Και αυτό μπορεί να είναι σε ορισμένε ε, περιπτώσει αυτό να είναι σωστό, αλλά για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το ζήτημα του μεταναστευτικού και των προσφύγων, συχνά δεν βλέπουν να υπάρχει απαραίτητη αλληλεγγύη. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο, ο Γιον Λάιλεν τώρα. Ευχαριστώ την Επιτροπή των Περιφερειών και την εξαιρετική ε, γνωμοδότηση από τη δική της ε, πλευρά. Ουσιαστικά αποτελεί το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στην επόμενη ε, στο επόμενο κοινοβούλιο, δηλαδή το πώς μπορούμε να επιτύχουμε και να συνδιαμορφώσουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία ε, ε, ανάμεσα στις θέσεις που προσβεύουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών. Ε, σίγουρα η Ευρώπη δεν είναι η Βρυξέλλες. Η Ευρώπη είμαστε όλοι εμείς, ανεξαρτήτως του που κατοικούμε. Και ακριβώς το ζητούμενο είναι αυτό, να το καταδείξουμε αυτό στους πολίτες μας, να το καταστήσουμε σαφές και να απηχείται αυτό και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεών μας. Ε, το δικαστήριο μία φορά είχε εκδώσει μία απόφαση σε ό,τι αφορά ε, την ε, διαδικασία ενσωμάτωση αυτών των διαδικασιών των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και η ίδια υποχρέωση νομίζω βαρύνει και τις αρχές και τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκηση. το γνωρίζει καλά αυτό η Επιτροπή των Περιφερειών. Εγώ είχα εργαστεί για πέντε χρόνια εκεί και είδα πώς ακριβώς λαμβάνει υπόψη της ε, τον ρόλο των, ε, των πόλεων και των περιφερειών σε αυτή τη διαδικασία. Ε, νομίζω πως ε, είναι πολύ σημαντικό αυτή η διάσταση να ενσωματωθεί στο μέλλον και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θεωρώ πως είναι πραγματικά σημαντικό γιατί το ε, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αποτελεί τη βασική κατευθυντήρια γραμμή, αν θέλετε, το βασικό άξονα στον οποίο κινείται η ευρωπαϊκή πολιτική. Επίσης, καταφέραμε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το δύσκολο ζήτημα της μετανάστευσης να εξασφαλίσουμε μια γραμμή του προπολογισμού, ειδικότερα ακριβώ για του Δήμου και τι ε, κοινότητε. Δηλαδή, όποιο κάνει κάτι ε, με δική του πρωτοβουλία θα πρέπει να ανταμείβεται γι' αυτό. Θεωρώ πω ε, πραγματικά να το, να το χειροκροτήσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν διάφορα επίπεδα βέβαια τα οποία διακυβέρνηση τα οποία διακείται αρνητικά απέναντι στη μετανάστευση. και βέβαια και στο επίπεδο της εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μόνο σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι εφικτή αυτή η υλοποίηση. Και σωστά ανέφερε και η κυρία Ρή ότι η κοινωνική διάσταση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τονιστεί περισσότερο ε, στην ε, επόμενη βουλευτική θητεία. Δηλαδή η ενιαία αγορά είναι ένα ψυχρό εντό εισαγωγικών ε, προϊόν. Δηλαδή δεν ζουν μόνο από την εργασία τους και ως καταναλωτές οι πολίτε μα. Ε, και νομίζω ε, πως είναι μια καλή ιδέα η θεσμοθέτηση αυτού του, του διαλόγου που ανέφερε η συνάδελφος. Δηλαδή, ο διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να είναι μόνιμος, όχι μόνο εν ώψη ευρωπαϊκών ε, εκλογών. Και ίσως θα μπορούσαμε να περιλάβουμε και ένα τμήμα ακρόαση σε αυτό το πλαίσιο αυτού του διαλόγου, δηλαδή να αφουγκραστούμε τους δικούς μας πολίτες για να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα και από την πλευρά των σοσιαλδημοκρατών πραγματικά ε, δεχτούμεθα πολύ θετικά απέναντι σε μια επικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών. Ευχαριστώ κύριο Σεροπέτο Τσάντη. Καλημέρα. Καλημέρα από την Σέρβον Πολιτική Ομάδα. Θέλω να έχουμε μια διακυβέρνηση πιο ισχυρή ε, από την βάση προς την ε, κορυφή. και το ίδιο να ισχύει όσον αφορά το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί δεν θέλουμε να είναι μόνο τοπικέ αρχέ ε, φορεί που πρέπει κάποιε φορέ να του ε, ε, συμβουλευόμαστε. Θέλουμε η επικουρικότητα να εφαρμόζεται πιο σωστά και έτσι να μπορούμε να έχουμε μια διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα και να γίνεται αυτό όποτε χρειάζεται και οι πόλεις οι δήμοι, οι κοινότητε, οι περιφέρειες να, όταν πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα, όταν να έχουν τη δυνατότητα να αυτοδιακυβερνηθούν. Οπότε έχουμε την task για την ε, επικουρικότητα που καταλήγει στο ότι θα πρέπει να είναι ενεργή, ε, δυναμική η επικουρικότητα και έτσι να μπορούν ε, δήμοι, κοινότητε, περιφέρειες να συμμετάσχουν στο νομοθετικό γίγνεσθε και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει περισσότερη συνέπεια, να υπάρχει περισσότερη αναλογικότητα και επικουρικότητα, οπότε ε, να μην είναι η νομοθεσία ε, περίπλοκη και να είναι πιο εύκολο να υλοποιηθεί, να εφαρμοστεί και να βοηθηθούν έτσι οι τοπικές αρχές και οι περιφερειακές αρχές. Αν έρχεται η ώρα της εφαρμογής του κοινωτικού δικαίου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη ε, των περιφερειών και αυτό θα πρέπει να διέπει την σταγματική λειτουργία της Ένωσης να έχουμε περισσότερο σημαντικό ρόλο και να συμμετέχουμε περισσότερο στην διαδικασία λήψης αποβάσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι θα κερδίσουμε πάλι την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων. Εμείς, οι εκπρόσωποι του κόσμου από εκείνο το επίπεδο, κάθε μέρα έρχονται στο γραφείο μας οι, Ευρωπαίοι και μας τα λένε. Ε, αυτό θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και επομένω γι' αυτό θα πρέπει να συμμετέχουμε στην λήψη αποφάσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριος Τσαλιλόντι από τους φιλελευθέρους. Thank you for giving me... Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συμβάρω και εγώ στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Καθότι Ιρλανδός, λυπούμε για το Brexit. Όμως θέλω οι εναπομείνασε χώρε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπόλοιποι 27, να αξιοποιήσουν αυτή τη συγκυρία για τη βελτίωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι πρέπει να χαίρουν ε, τη ε, εσωτερική αγορά, τη ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όμω πάνω απ' όλα το κράτο δικαίου θα πρέπει να γίνεται σεβαστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω από το φω των όσων συμβαίνουν σε ορισμένα κατημέλη. Είναι σημαντικό για μα, ιδιαίτερα του Ιρλανδού, να μην υπάρχει ε, σύνορο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου και ελπίζω να ακολουθήσουμε αυτή την ε, άγουσα και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να ζητήσω από το Βρετανικό Συμβούλιο, Κοινοβούλιο να υιοθετήσει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών θα θέλαμε να συνεργαστούμε από κοινού ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο με μια νέα μορφή, γιατί έχουμε κοινέ προκλήσεις για τη μετανάστευση, για την ε, ανεργία, την ανασφάλεια, την κλιματική αλλαγή και απαιτείται μια συλλογική απάντηση. Όπως έχουν πει και άλλοι και θέλω και εγώ να επαναλάβω, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ακολουθεί την κατάλληλη προσέγγιση ανάλογα με το θέμα. Πιο ευρωπαϊκή, πιο εθνική. Και είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα για να πετύχουμε τους κοινού μα στόχου Στην Ιρλανδία, όταν μιλούμε για το μέλλον της Ευρώπης, λέμε το μέλλον είναι η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you uh, very much for the... Ευχαριστούμε πολύ. Από τους Πρασίνους, ο κύριος Γιουκάναν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Που μου δίνετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η γνωμοδότηση τη Επιτροπή των Περιφερειών για το μέλλον τη Ευρώπη είναι ένα εξαιρετικό έγγραφο. Αποτελεί όμω μόλι την αφετηρία, γιατί μπαίνει στην ουσία που είναι η τοπική και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ε, που βρίσκονται πιο κοντά στου πολίτε μα και μας έχουν εκλέξει για να μεταφέρουμε τις απόψεις και γνώμες τους. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός αυτό το χάσμα που υπάρχει μεταξύ ευρωπαϊκού και τοπικού επίπεδου φαίνεται και από το πόσο λίγο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μα για αυτό το ζήτημα. Όπω ακούτε την πληροφορά μου, είμαι Σκοτσέζο και στη Σκοτία όλοι οι φορεί τη τοπική αυτοδιοίκησης έχουν ψηφίσει για την παραμονή τους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη δική μου εκλογική περιφέρεια ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό υπέρ της παραμονής και αυτό επειδή εμείς εξηγήσαμε τα ωφέλη ε, της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γίνεται με πολλές μορφές, ε, όταν έχουμε δημόσια έργα, όταν έχουμε ε, άλλες μορφές ε, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Πάντα προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι όλα αυτά προκύπτουν από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται άμεσα με την καθημερινότητά μας. και ε, μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα ότι δεν χρειάζεται κανείς να χάσει την ταυτότητά του που ε, σε μεγάλο βαθμό ήταν και ο λόγος που ψήφισαν ε, πολλοί στον Ηνωμένο Βασίλειο για την αποχώρηση, γιατί φοβήθηκαν ότι θα χάσουν την ταυτότητά τους. Δεν χρειάζεται κανείς να χάσει την ταυτότητά του. Κάθε περιοχή όμως πρέπει να διασφαλίσει ότι ο πληθυσμός δεν θα νιώσει διάκριση εναντίον του. Και πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να αλλάξει ως προς αυτό, να ακούγονται όλες αυτές οι φωνές, να δίνονται αυτές οι ευκαιρίες. Πολλοί θα πούν ακριβώς τα ίδια, πολλοί θα προέρχονται από τις ίδιες ακριβώς περιοχές, όμως πρέπει να νιώσουν ότι κάποιος τους ακούει. Μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Εξετάζουμε όλους τους τομείς, ε, την ενσωμάτωση, τη συμπερίληψη, εμείς έχουμε ένα κοινό έχουμε δύο σχολεία, ένα καθολικό και ένα εβραϊκό, που συστεγάζονται. Και στα δύο συμμετέχει σημαντικό μουσουλμανικό στοιχείο, πολλοί μαθητές. Επομένω, εκεί ακριβώς αντιμετωπίζουμε ε, το θέμα της συμπερίληψης και της ε, κοινωνικής ένταξης. Τα πράγματα δεν θα αλλάξουν βέβαια από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι σημαντικό όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια φωνή το μέλλον είναι η νεολαία μας. Εμείς ψηφίσαμε να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σκωτία. Θα ακολουθήσουμε τον δρόμο που ε, ελπίζουμε να μας φέρει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί ξέρουμε ότι το μέλλον μας είναι κοινό, χωρίς να χάσουμε τα ταυτότητά μας, ξέρουμε ότι από κοινού όμως μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Από την άλλη βέβαια, εγώ είμαι και υπέρ τη ε, σκοτσέζικης ανεξαρτησίας, αλλά ε, έχουμε κοινέ αρμοδιότητες και συνεργαζόμαστε με τις αρχές. Μπορούμε να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα. Να συνεργαστούμε εκεί που μπορούμε προς όφελος ε, των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εσπυρίδων έχει ζητήσει το λόγο εξ ονόματος του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Λίγε λίγες μέρες πριν η Ευρώπη γιόρτασε την επέτειο των 100 χρόνων από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέσα από τις τάχτες των δύο παγκοσμίων πολέμων, οραματιστές και αποφασισμένοι ηγέτες, στο όνομα των προσδοκιών των ευρωπαϊκών λαών, οικοδόμησαν την Ευρώπη της ειρήνης, της δημοκρατίας, της σταθερότητας και της προόδου. Τις μέρες μας, ωστόσο, οι αρχές αυτές παραγνωρίζονται. Επικίνδυνες δυνάμεις που υπηρετούν τον λαϊκισμό τον εθνικισμό, αποδυναμώνει το περιεχόμενο της Ευρώπης, εκμεταλλευόμενα στην οικονομική κρίση, τη ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών και κυρίως την ανασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών που καλλιεργούν διαδοχικές τρομοκρατικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια. Το, το ευρωπαϊκό επιχείρημα αμφισβητείται. Τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλονίζονται και για πρώτη φορά στην ιστορία της με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου γίνεται μικρότερη. Επιτεύγματα όπως η πλέον μακροχρόνια ειρήνη στην ιστορία της Ευρώπης, η διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αξιών, η πολιτική ελευθερία, η ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, ιδεών, κεφαλαίων και τόσα άλλα επιτεύγματα θεωρούνται δεδομένα κυρίως από τις νεότερες γενιές. Από την άλλη πλευρά, η ενιαία αγορά από μόνη της δεν μπορεί πλέον να συνιστά το όραμα για τους νέους και τη συνοχή της Ευρώπης. Απαιτούνται άμεσα γενναίε πολιτικέ που θα υπαγορεύονται από την αρχή τη αλληλεγγύη και τη υπευθυνότητα και θα στοχεύουν στην οικονομική, εδαφική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σύγκληση του βιωτικού επίπεδου όλων των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κύρος της μεγάλη μα οικογένεια έναντι των άλλων χωρών πρέπει να ενισχυθεί με τη δημιουργία κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή άμυνα και κανόνων που αφορούν την οικονομία. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί ή να μην πρέπει να γίνει μια ομοσπονδιακή ένωση όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής, μπορεί όμως να αποκτήσει ομοσπονδιακού τύπου λειτουργίες στους τομείς εκείνους που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστούν όλα εκείνα που προϋποθέτουν την ασφάλεια, την ευημερία και το κοινό μέλλον των πολιτών μας. Ισχυρή ίσον ενωμένη και ενωμένη ίσον περισσότερη Ευρώπη με ό,τι αυτό σημαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, you, George um, Ευχαριστώ. του Έλκα να σας καλωσορίσουμε σε αυτήν την τόσο σημαντική συζήτηση και θέλω τώρα να εστιάσουμε την προσοχή μας στο εξή. Θα μπορούσαμε να το πούμε πρόβλημα των πολιτών, αλλά τελικά, ναι. Υπάρχει υποστήριξη προς την Ευρώπη, αλλά δεν έχω πιστεί ότι αυτή η υποστήριξη αναγκαστικά αφορά τις ε, σημερινές ε, ρυθμίσεις, το ε, θεσμικό καθεστώς που διέπει την Ευρώπη, που είναι δυσκίνητο, δεν έχει ευέλιξη. Δύσκολο να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό, αλλά η συνέπεια είναι ότι δεν υπάρχει ταύτιση με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι τώρα. Και αυτούς και για τον περισσότερο κόσμο. Ναι, να έχουμε δημοκρατική Ευρώπη. Αλλά το θέμα είναι ε, υπάρχει ένα, ένα κενό όσον αφορά το γιατί θέλουμε την ολοκλήρωση και το θέμα είναι το πού πήραμε το λάθος δρόμο. Είναι το θέμα το ποιες είναι αυτές οι αξίες. Ε, αναδεικνύουμε τις αξίες που εμάς ε, καθορίζουν, αλλά όχι αυτά που θέλει ο κόσμος. Γκράς. Και μετά εσείς κύρια κυρία Μαγκέρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας παραπέμπω σε αυτό που είπε ο πρώτος Λάμπερτς για την ενσάρκωση του κακού. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την τόσο αρνητική άποψη για την Ευρώπη. Εγώ προέρχομαι από μια μικρή χώρα, από το Λουξεμβούργο. Βέβαια, έχουμε μακρά φιλοευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή παράδοση. Και όλοι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτούς που θέλουν λιγότερη Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει να προβληματιστούμε μήπως θα πρέπει στη χώρα μας να έχουμε μια καινούργια γιορτή ε, ως επέτειο, ας πούμε 9 Μαρτίου με συμβολική αξία και σε όλες τις χώρες να γίνεται με κάποια συζήτηση να είναι κάτι ως σύμβολο και έτσι όλοι που ενδιαφέρονται για την Ευρώπη αλλά και όλοι που δυσπιστούν χρειάζεται επομένως περισσότερη προσπάθεια και η Επιτροπή των Περιφερειών έχει ρόλο να διαδραματίσει σε κάθε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό. Α, πολύ αξιόλογο αυτό που οργανώσατε σήμερα το πρωί αυτή την συζήτησή μας. Μπράβο. Όλοι όλοι οι αιρετοί έχουν ρόλο σημαντικό να διαδραματίσουν στο μέλλον, άρα θα πρέπει να κάνουμε παραπάνω προσπάθεια και να πείσουμε κυρίως εκείνους που ακόμα έχουν την επιφύλαξη ότι η Ευρώπη δεν είναι η λύση για το μέλλον. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι μόνο η Ευρώπη είναι η λύση για το μέλλον και θα πρέπει να δώσουμε μαζί τον αγώνα για την επιτυχία του στόχου. Κύριε Μαγιάρα. Θα είμαι σύντομη και θέλω να συγχαρώ τον κύριο Σεφλίν για την πρωτοβουλία του όσον αφορά τους πολίτες. Ναι, χρειάζεται η Ευρώπη, Ευρώπη των πολιτών. Μου αρέσει να λέω όχι περισσότερη Ευρώπη, καλύτερη Ευρώπη. Ε... Εμείς ευχαριστούμε, λέει η πρόεδρος. Λάιναν. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να αναφέρω ότι οι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατοχυρωμένε ε, στι συνθήκε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια όλα τα κράτη-μέλη τα οποία υπέγραψαν αυτέ τι συνθήκε, έχουν δεσμευτεί. Δεν μπορούν ε, δηλαδή να αποφασίζουν εκ των υστέρων ότι θέλουν να αποκλίνουν ε, είτε σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου, είτε σε ό,τι αφορά το δημοκρατικό σύνταγμα, είτε σε ό,τι αφορά τον πλουραλισμό ή την ελευθερία σε ό,τι αφορά την έρευνα και ούτω Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να επιλέγουμε ο καθένας ε, τι είναι σωστό και τι είναι λάθος ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το κάνουμε αυτό θα καταρρεύσει το οικοδόμημα. Έχουμε συμφωνήσει επί κοινών αξιών στο υψηλότερο ε, δυνατό επίπεδο, οπότε όλοι δεσμεύονται από τις ίδιες αξίες. Σε αυτό βασίζεται και ο πλουραλισμός, ότι δηλαδή η πολυμερής προσέγγιση, ότι δηλαδή αν συμφωνούμε επί κάποιων αξιών, τότε θα πρέπει να μας δεσμεύουν όλους. Ο Καλχάνης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ενέπνευσαν ιδιαίτερα τα σχόλια των συναδέλφων. Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρούν ότι θα πρέπει να εντείνουμε και να τελειοποιήσουμε έτσι περαιτέρω τις ε, σχέσεις μεταξύ των δύο θεσμικών μας οργάνων. Και εγώ συμμερίζομαι αυτή την πεποίθηση Έχουμε ένα σαφή στόχο, στρατηγικό στόχο, μέσω της ε, εκπόνησης ε, εκθέσεων της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς εμείς εκπροσωπούμε την τοπική αυτοδιοίκηση και έτσι λαμβάνουμε και σας τροφοδοτούμε με όλα τα στοιχεία που θέλουν να σας μεταφέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό είναι ο μηχανισμός ε, με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο σε αυτό το μονοπάτι. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε κατά νου την ε, τρομερή ε, πολυμορφία του θεσμικού πλαισίου στα επιμέρους κράτη-μέλη. Πράγματι, η αποκέντρωση, όπως θέλετε πείτε το, έχει να κάνει ε, και είναι θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας κάθε κράτος μέλους. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα έχει όλα αυτά κατά νου, αλλά η πολυμορφία του τοπικού και περιφερειακού τοπίου ε, μας ε, δείχνει ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε διαφορετικά επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ η Επιτροπή μας με κάθε τα ταπεινοφροσύνη μπορώ να σα πω ότι διαδραματίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, γιατί ούτε οι ευρωβουλευτέ, ούτε ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε κανένα άλλο μπορεί να μιλήσει με 1.500 δημάρχου ε, στην Ευρώπη κάθε μέρα. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος μας λοιπόν. Μετά, δύο ακόμα πράγματα. Αν θέλουμε να έχουμε πιο στενούς δεσμούς με τους πολίτες μας, πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τους διάβλους επικοινωνίας. Μονίμως δηλαδή να υπάρχει, να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός, αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και τώρα πρέπει να βρούμε από τεχνική άποψη ε, τον τρόπο να ελοποιηθεί αυτό όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Και φυσικά και πρέπει να υποβάλουμε προτάσεις ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Και η τελευταία μου παρατήρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μέλλον μας. Όμως δεν αρκεί να το πιστεύουν αυτό οι πολιτικοί. Πρέπει να πείσουμε και τους πολίτες. Και αυτό γίνεται μέσω μιας διαδραστικής διαδικασίας. Που εντάσσεται σε αυτή την ε, περιβόητη συζήτηση ευρωπαϊκή ηθαγένεια έναντι εθνικής ταυτότητας, και παράλληλα βλέπουμε ότι περνάμε μια περίοδο που όλα αυτά δεν πηγαίνουν πολύ ομαλά και τα έχουμε ξανασυζητήσει. Το βασικό όμως είναι να κατανοήσουμε ότι τα τρία επίπεδα δεν ε, λειτουργούν διαζευτικά ή σε αντίθεση το ένα προς το άλλο, αλλά από κοινού. Οπότε το ευρωπαϊκό εγχείρημα ε, είναι η σύνθεση όλων των υπόλοιπων επιπέδων. Το ευρωπαϊκό δεν αντικαθιστά το τοπικό ή το περιφερειακό ή το εθνικό. Απλώς ε, αξιοποιεί περαιτέρω τα όσα κάνουμε για να έχουμε κοινά αποτελέσματα. Κάτι που ε, αντικατοπτρίζεται και στον κοινό μας στόχο και την πεποίθησή μας ότι το μέλλον μας είναι η Ευρώπη. Θέλει να πάρει η κυρία Ντούντεν το λόγο, παρότι σύντομα θα διακοπεί η διερμηνία. Παρακαλώ. No. No, okay. So I just like to we are approaching the end of our discussion. Ωραία, φτάσαμε στο τέλος ε, της ε, σημερινής συζήτησης. Ελπίζω να είναι και η αρχή της συνέχειας. Πρέπει να προστατεύσετε και την Ευρώπη κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς ευρωεκλογών με πολλούς κινδύνους μπροστά μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως και για αυτή τη γνωμοδότηση, γιατί ε, ανέφερε και συγκεκριμένα σημεία προβληματισμού και ε, τη δυσαρέσκεια που υπάρχει. Και εμείς τα ξέρουμε ότι δεν είναι όλα όπως πρέπει, αλλά είναι μια διαδικασία εν εξελίξη και αυτή είναι και η ευθύνη όλων εμάς των ερετών εκπροσώπων. Για τους συναδέλφους που μίλησαν για το Brexit, σύντομα θα περάσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συμφωνία. Ελπίζουμε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή λύση, μια έξοδος δυνάμει μιας ε, καλής συμφωνίας, για να αποφύγουμε δραματικές καταστάσεις ε, απουσία συμφωνίας. Και στο Κοινοβούλιο πραγματικά νιώσαμε ότι έπρεπε να είμαστε επικοδομητικά θετική. Παρότι λυπούμεθα λοιπόν για την αποχώρηση των Βρετανών, σεβόμαστε τα όσα κάνουν, τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, να δοθεί ένα αίσιο τέλος σε αυτή την ε, αμοιβαία επιζήμια βέβαια διαδικασία. Όμως ε, και η Βρετανική πλευρά έχει δραματίσει σημαντικό ρόλο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ελπίζω να συνεχιστεί ε, αυτή η συνεργασία και στην επόμενη θητεία. Καλή συνέχεια.